May I ask you, colleagues, to take seat? I will give a couple of minutes uh, during. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγα λεπτά στην υποψηφία επίτροπο αλλά και στους δημοσιογράφους για να πάρουν τις φωτογραφίες και μετά θα τους ζητήσω να φύγουν από την αίθουσα ή μάλλον να καθίσουν κάπου αλλού. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Να σας καλωσορίσω κύριε Βέσταγκερ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Είναι η τρίτη ακρόαση που διοργανώνει η Επίτροπη ΕΚΟΝ. Έχουμε γίνει μηχανή ακροάσεων, αλλά είναι μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε λοιπόν τους προτινομένους επιτρόπους και στο σύνολό τους και μεμονωμένα επί τη βάση των αρμοδιοτήτων τους, της ευρωπαϊκής τους αφοσίωσης και της ανεξαρτησίας τους της προσωπικής από διάφορα συμφέροντα και φυσικά να αξιολογήσουμε και τις πολιτικές τους προτεραιότητες και τη δυνατότητα συνεισφοράς τους στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κανόνες μας είναι οι εξής. Η υποψηφία επίτροπος θα κληθεί να κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση 15 λεπτών το πολύ. Και αμέσως μετά θα υπάρξουν 45 ερωτήσεις, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. και στο τέλος θα υπάρξουν ε, ομιλίες από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων. Θα ζητήσω από όλους τους ομιλητές παρακαλώ να σεβαστούν το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Ένα λεπτό και μετά δύο λεπτά όπως είπα η απάντηση. Η διευμηνία παρέχεται σε 23 γλώσσες. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω και από τους ομιλητές παρακαλώ να μην ομιλείτε πάρα πολύ γρήγορα και να σας διαβεβαιώσω ότι η συζήτηση αυτή θα μεταδοθεί από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στην υποψηφία επίτροπο, να πω ότι εμείς ε, προωθούμε σαν στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Είναι ένας ιστορικός στόχος αν θέλετε και έχει πολλές αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τις δυνατότητες αυτές και στο, στο βαθμό του εφικτού βέβαια κάθε φορά να μπορέσουμε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση τη σωστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η λειτουργική μορφή του ανταγωνισμού σε τομείς όπως τα χρηματοπιστωτικά και οι νέες τεχνολογίες θα συνεισφέρει τα μάλα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε όπως το θέμα των κρατικών μονοπωλίων, τα προβλήματα του πιστοτικού τομέα και ο ενιαίος μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαγκρέτε Βέισταγκερ για την παρουσίασή της. Κύριε Πρόεδρε Γουαλτιέρη. Α, ωραία, όλα εντάξει, ναι. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. είναι πράγματι μια ευκαιρία για μένα να εκφράσω την ε, πολιτική μου, τα πολιτικά μου κίνητρα για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την ακρόαση αυτή. Μας ενδιαφέρει όλους να μπορέσουν όλα τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθούν σε ισορροπία με τη φύση τους. Θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται μέσα σε μια οικονομία η οποία είναι βιώσιμη και δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι απόκληροι. Μια ανοιχτή κοινωνία, μια κοινωνία η οποία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, αν με επικυρώσετε ως, ε, υποψή, ως, επί, ως επίτροπο, θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έχω κάνει σε όλη μου την πολιτική καριέρα. Να συμβάλλω, ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν εξουσία να μην μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να επιβληθούν στους μικρούς. Στους μικρούς. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να μην υπάρχουν άτομα τα οποία αποκλείονται από την κοινωνία ή είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης. Με έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι θεμητός και ισοδίκαιος μπορούν όλες οι ιδέες να ανθίσουν. Όλοι οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία της επιλογής σε ε, προσιτές τιμές. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μπορώ να έλθω ενώπιον της Επιτροπής σας. Για πρώτη φορά ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 25 χρόνια. Ποτέ μου όμως δεν είχα φανταστεί ότι σήμερα θα βρεθώ ενώπιον σας και φυσικά είναι μια μεγάλη τιμή για μένα και την αντιμετωπίζω με μεγάλη ταπεινοφροσύνη αυτή την τιμή. Ήμουν 21 ετών όταν μπήκα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του πολιτικού μου στη Δανία. Το σύνθημα με το οποίο κάναμε εκστρατεία ήταν «Πιστεύουμε στην Ευρώπη». Και εγώ πιστεύω πράγματι στην Ευρώπη. Προχωρούμε τώρα, αν γυρίσω τρία χρόνια πίσω από σήμερα, σχεδόν ακριβώς τρία χρόνια, έγινα υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Εσωτερικών στη χώρα μου και πήγα στην πρώτη μου συνεδρίαση του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Ήταν μια χρονική στιγμή μεγάλης αβεβαιότητας και είδα στο Συμβούλιο και ένιωσα πως η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να γίνει μια σειρά συγκεκριμένων και πρακτικών λύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ξεπεράσαμε την θύαλα της κρίσης ήταν με την αλληλεγγύη μεταξύ μας με το να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε οι μεν στους δε και με το να εργαστούμε για το κοινό συμφέρον. Αυτό ήταν το πνεύμα το οποίο επικράτησε στο Συμβουλιακό ΦΙΝ. Χάρη και στις σόφρονες αποφάσεις που πήρε η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, μπορέσαμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης. Ξεκινώ με αυτές τις αναμνήσεις, γιατί θέλω να μεταφέρω το ίδιο πνεύμα στην θέση στο αξίωμα αυτό για το οποίο είμαι υποψήφια σήμερα ενώπιόν σας. Πιστεύω ότι η προάσπιση του κοινού συμφέροντος πρέπει να είναι και ο ακρογωνίος λίθος μιας πολιτικής ανταγωνισμού. Δεν είμαι συνηθισμένη να λέω μεγάλα λόγια. Πιστεύω όμως ότι εδώ είναι πράγματι περί αυτού που πρόκειται όταν δείτε πόσο σημαντικές είναι οι εξουσίες, οι εκτελεστικές εξουσίες που έχει η Κομισιόν στον τομέα του ανταγωνισμού. Η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η αυστηρότητα για να εξασφαλίσουμε το κράτος δικαίου είναι απαραίτητες. Η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά την οικονομική φιλοσοφία, σε ό,τι αφορά τον νόμο. Αυτή θα είναι και η βάση για την προσωπική μου δράση. Θα είμαι ανοιχτή να ακούσω τις απόψεις όλων από τις μεγαλύτερες πολιτικές εταιρείε μέχρι τους εκπροσώπους μικρών εταιρεών. Από τα κράτη, μέλη, μέχρι τους απλούς πολίτες. Αλλά η ανάλυση του προσωπικού μου και η δική μου τελική κρίση δεν θα παρασύρεται από τις απόψεις κανενός. Το κύρος της πολιτικής ανταγωνισμού και της εφαρμογής της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεξαρτησία μας, στην αμεροληψία μας και επίσης και στο σεβασμό της εμπιστευτικότητας στην αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων. Εάν με επικυρώσετε ως Επίτροπο, θα υπερασπιστώ αυτή την παράδοση αόπνος. Οι έρευνες θα γίνονται και οι αποφάσεις θα προτείνονται στο Σώμα των Επιτρόπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, από την ισχύ ή το μέγεθος μιας εταιρείας και σε περιπτώσεις κρατικής βοήθειας ανεξάρτητα από τις εμπλεκόμενες χώρες. Για μένα αυτές είναι οι κέρδιες αξίες της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού. Μεταξύ των πολλών πραγμάτων που θαυμάζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η δική σας προσήλωση σε αυτές ακριβώς τις αξίες. Εάν εγκριθώ από εσά, προσβλέπω να εργαστώ μαζί σας, να συνεργαστώ μαζί σας για να εξασφαλίσω ότι ακριβώς η αμεροληψία η ουδετερότητα και η αυστηρότητα θα είναι οι οδηγές αρχές για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Όπως σας είπα προηγουμένως, η οικονομική κρίση καταφέραμε να περιορίσουμε τις αρνητικές πτυχές της. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νιώσει την ύφεση, αυξανόμενη, την αυξανόμενη ένδια και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Έχουμε ενώπιόν μας μια σαφή πρόκληση. Να επαναφέρουμε την Ευρώπη στα πόδια της, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης, να είμαστε καινοτόμοι, να ξαναφέρουμε μια δυναμική και κοινωνική συνοχή. Η πολιτική ανταγωνισμού έχει να διαδραματίσει ένα κέριο ρόλο στο να υποστηρίξει την έκκληση του Πρόεδρου της Κομισιόν για να υπάρξει μια ανάκαμψη σε επίπεδο απασχόλησης, μεγένθησης και επένδυση για να αντιμετωπιστούν οι συνολικέ προκλήσει για τη βιομηχανία μα, για τι μικρέ και τι μεγάλε επιχειρήσει. Ο βασικό μου στόχο λοιπόν θα ήταν να αντιμετωπίσω τα κέρια εμπόδια για την ανάπτυξη και την καινοτομία που είναι απαραίτητη για τι θέσει απασχόληση. Οι επιτυχίε των εταιριών προκύπτουν από τον θεμητό ανταγωνισμό. Σε σημαντικέ αγορέ όμω, όπω είναι η ενεργειακή και η ψηφιακή αγορά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να εξασφαλίσουμε ότι οι κυρίαρχες εταιρείε σέβονται του κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και καινοτομία από μικρότερες και μεσαίες εταιρείε. Στον τομέα των κρατικών επιδοτήσεων θα ακολουθήσω το θεματολόγιο της, του εξυγχρονισμού των κρατικών αρρωγών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν όλα τα κρατημέλη να αναλάβουν όλο και περισσότερη ενεργή ευθύνη για τις ε, κρατικές επιδοτήσεις. Θα αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η διαφάνεια και ο ανοιχτό χαρακτήρας και θα μπορέσει και το κοινό να καταλάβει πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι σπάνιοι εθνικοί πόροι. Οι πολίτες θα έχουν μια σαφέστερη εικόνα του πώς χρησιμοποιούνται τα λεφτά των φορολογμένων. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μπορούν να είναι τμήμα μιας ευρύτερης συζήτησης. Ενίοτε η εφαρμογή των κρατικών αρρωγών και των κανόνων για τις συγχωνεύσεις και την ε, νομοθεσία αντιτράστ έχουν κάποιο βραχυχρόνιο, βραχυπρόθεσμο τίμημα. Ο θεμητός ανταγωνισμός και η αλλαγή στις αγορές μας έχουν εν καιρό ένα πραγματικό μέρισμα ανάπτυξης. Ένα πραγματικό μέρισμα, αλλά μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να έχουν κοινωνικό κόστος. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης για να εξασφαλίσω ότι οι παρεμβάσεις τους δεν αναχαιτίζουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Και συγχρόνως θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να εξασφαλίσω ότι τα συνοδευτικά μέτρα για αυτές τις μεταβάσεις λαμβάνουν πάντα υπόψη την κοινωνική διάσταση. Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε εδρεωμένες και υγιείς αρχές. Οι αρχές αυτές είναι σαφείς μέσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δοκιμαστεί από τον χρόνο. Το να κρατήσουμε την ενιαία αγορά ανοιχτή και να εξασφαλίσουμε ισότητα ανταγωνισμού, αυτή είναι η πιο άμεση στόχη της πολιτικής ανταγωνισμού. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πετύχουμε με τον τρόπο αυτό είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό από τον ίδιο τον ανταγωνισμό. Το στόχο της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. Από τότε που υπήρξε η πρώτη διατύπωση των κανόνων ανταγωνισμού στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ήδη λίγο που σας λέω. Η οικονομία μας είναι τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ψηφιακή οικονομία. Αυτή η εξέλιξη και άλλες εξελίξεις μας φέρνουν ενώπιον της πρόκλησης να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των αγορών για να μπορούμε να τις παρακολουθούμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ακονισμένα τα εργαλεία μας και να μπορέσουμε να προβλέπουμε τις αλλαγές στην οικονομία μας. Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο η πολιτική ανταγωνισμού παίζει ένα κέριο ρόλο για να μας βοηθήσει να έχουμε και πάλι οικονομική ανάπτυξη. Για μένα δεν είναι θέμα που αφορά μονάχα τις εταιρείε και τους καταναλωτές. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με τους πολίτες, με τους ανθρώπους, με εμάς τους ίδιους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι μικρές και οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να ανταγωνιστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η πειθαρχία των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας να είναι καινοτόμε και να ενισχυθούν. Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την πολιτική ανταγωνισμού όπως χρειαζόμαστε την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις επενδύσεις, το κεφάλαιο και μια καταρτισμένη εργασιακή δύναμη. Δεν είναι μια υγιής βιομηχανική πολιτική το να προστατεύουμε εταιρείε από τον ανταγωνισμό, γιατί αυτό είναι σε βάρος των ίδιων των καταναλωτών. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι το χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού έχει μοναχικό χαρακτήρα. Κάθε άλλο. Η καλύτερη ρύθμιση δημιουργεί και υποστηρίζει την ενιαία αγορά και παροτρύνει τις εταιρείες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η ρύθμιση δημιουργεί πραγματικότητε στον τομέα τη αγορά. Το είδαμε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου είχαν μείνει εθνικέ και κατακαιρματισμένε οι αγορέ για πολλά χρόνια μετά την αρχική φιλελευθερωποίηση. Λένε ορισμένοι ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μια πραγματική πολιτική ανταγωνισμού όταν δεν υπάρχει πραγματική επαγρύπνηση των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαφωνώ. Ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό ανταγωνισμό είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα συνεργαστώ και με του άλλου επιτρόπους. Είναι ένα από του λόγου για αυτό για, που ο ανταγωνισμό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ω ένα μοναχικό χαρτοφυλάκιο. Θέλω να συνεργαστώ και με εσά, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και άλλων επιτροπών Θέλω όμως και σε επίσημο και σε ανεπίσημο επίπεδο να συνεργαστώ μαζί σας. Ο καθένας σας ξέρει τη δική του εκλογική περιφέρεια πολύ καλύτερα, ξέρει τις ελπίδες και τις ανησυχίες των πολιτών του καλύτερα από όλους τους άλλους. Χρειάζεται να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις εκεί που είναι απαραίτητο να υπάρξουν ευρωπαϊκού επίπεδου λύσεις. Για να το κάνουμε αυτό, και παραθέτω αυτά που είπε ο πρόεδρο Γιούγκερ, πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και πιο φιλόδοξοι για τα μεγάλα πράγματα και πιο ταπεινοί και πιο μικροί για τα μικρά πράγματα. Ο συγχρονισμός <clears throat> των κρατικών επιδοτήσεων μα έχει θέσει στη σωστή τροχιά και μα βοηθάει να δούμε πού χρειάζονται οι παρεμβάσει μα ενώ συγχρόνω, βασιζόμαστε στα κατημέρια να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν καλύτερα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τραστ, θα πρέπει να εστιάσουμε στις επιχειρηματικές πρακτικές σε κέριου τομείς. Εγώ υποστηρίζω τον στεναρό ανταγωνισμό και δεν θέλω να εμποδίσω τις μεγάλες εταιρείε από το να ανταγωνίζονται σε επίπεδο ισότητας. Δεν θα διστάσω όμως να αμφισβητήσω τη δραστηριότητα μεγάλων εταιριών όταν με καταχρηστικό τρόπο θέλουν να πιέσουν τους μικρότερους παίκτες από την αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι τις ίδιες αξίες υποστηρίζετε και εσείς. Γιατί η πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι μία μορφή γραφειοκρατίας. Ακολουθεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υποστηρίζω, θα, ελπίζω θα έχω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν με επικυρώσετε θα συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας και φυσικά θα είμαι προσιλωμένη σε ένα τακτικό διάλογο στα πλαίσια του ομοιβαίου σεβασμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Όχι μόνο αυτό είναι επίσημα απαραίτητο, αλλά όταν είναι δυνατό. Είναι προς το συμφέρον των πολιτών και επομένως και προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους εκφράζει και τους αντιπροσωπεύει. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό ξεκινάμε μια ανοιχτή, έντονη και καρποφόρα εταιρική σχέση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Ο πρώτος είναι ο Μπούρκα Μπάλτς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Βεστάκερ. Το ερώτημα μου έχει να κάνει με την διεθνοποίηση του ανταγωνισμού. Προβλέπετε ότι του χρόνου το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης έως και το 90% θα λαμβάνει χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικές μας επιχειρήσεις χάνουν τον αγώνα δρόμα, δρόμου της παγκοσμιοποίησης και μείνουν πίσω. Χρειάζεται να προωθηθούν στρατηγική σημασία τομείς όπως ε, η αεροβιομηχανία, όπως η κατασκευαστική, όπως οι τηλεπικοινωνίες. Ε, ερωτώ λοιπόν εάν θεωρείτε ότι η τωρινή πολιτική ανταγωνισμού όπως έχει χαραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει τους, τις προκλήσεις παγκοσμιοποίησης και των μεγάλων αυτών προκλήσεων. Και μια δεύτερη ερώτηση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού και κυρίως όταν αναφερόμαστε σε στρατηγικά στρατηγικούς κλάδους της βιομηχανίας ε, δεν θα πρέπει να έχουν κάποια ευκαιρία για να ε, επιβιώσουν στον αγώνα αυτό στο διεθνές σκηνικό. Τι είδους μέσα βλέπετε για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Απάντηση. Ακριβώς αυτό είναι και στο επίκεντρο των πολλών, ανησυχιών πολλών πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ότι όπου και να δουλεύουν μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως οπουδήποτε αναπτύσσει δραστηριότητε της μια εταιρεία στην Ευρώπη, οι κανόνες να είναι οι ίδιοι, ανεξάρτητα του ποιος είναι ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, οπουδήποτε και να δουλεύει η επιχείρηση ε, θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες. Επίσης, θα πρέπει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα, να λέμε πότε διαπραγματευόμαστε για το εμπόριο και όποτε ε, συζητούμε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει να τα λέμε όλα ανοιχτά. Όπως λέμε στα δανέζικα και το μεταφράζουμε, ε, να είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Τα χαρτιά ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Για να είναι σαφείς οι όροι. Και ταυτόχρονα έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε το διεθνή ανταγωνισμό. Ε, βλέπω ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναπτύξει μια δραστηριότητα πεντάστερη υψηλής ποιότητας, την οποία όχι μόνο θα πρέπει να υποβαθμίσουμε, αλλά να πείσουμε και τους άλλους να αναπτύξουν καλύτερο επίπεδο για να βελτιωθεί το επίπεδο του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως υπάρχουν πολλά θέματα που θα πρέπει να δούμε ε, γιατί έχουμε και κρίσιμου τομεί όσον αφορά τα, πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα τη βιομηχανική ιδιοκτησία ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξω μαζί με του ε, συναδέλφου που έχουν παράλληλα χαρτοφυλάκια. Ευχαριστώ, Φερέιρα, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ, υποψήφια επίτροπε. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση για τι τράπεζε στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, από ό,τι ορίζει η οδηγία για την ε, διάσωση των τραπεζών, ε, μπορεί να χορηγηθεί ειδική υποστήριξη σε μια τράπεζα χωρίς να τεθεί σε κίνηση ο μηχανισμός, βοήθεια με Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωράει σε μια συνολική αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να προηγηθεί της νέας εποπτικής δραστηριότητας που θα αναλάβει. Βάσει αυτής της ασκήσεως, το μπορεί να χρειαστεί προσθήκη κεφαλαίου για μια τράπεζα. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα εξασφαλίσετε ότι οι δεσμεύσεις αυτές για την παροχή κεφαλαίου δεν θα θέσουν αμφιβόλο την ισότητα ανταγωνισμού ότι θα είναι συμβατές με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν θα χρησιμοποιηθούν για να κρατήσουν εν ζωή τράπεζες οι οποίες δεν είναι πια βιώσιμες. Ένα από τα πράγματα που του τους ανθρώπους είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας μετά από όλα τα δεινά που έχει προξενήσει και τις κρίσεις που έχει προκαλέσει όλα αυτά τα χρόνια και πώς θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι ακριβώς λόγω αυτής της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης εκφράζω αυτές τις ιδιαίτερες ε, ε, ε, ιδέες. Οι προκλήσεις της οδηγίας αυτής, της BLRD, δεν ε, έχουν τεθεί σε εφαρμογή ακόμα, δεν έχουν ε, δραστηριοποιηθεί ακόμα. Γιατί, για να μην κληθεί ο πολίτης να πληρώσει τα σπασμένα. Υπάρχουν άλλα στάδια ε, υποστήριξη των τραπεζών πριν φτάσει η ώρα να τεθεί σε λειτουργία η BLRD. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα από τη μία του bail out και από την άλλη του bail in αν βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μια τράπεζα. Θα έχω εγώ πολλή δουλειά μαζί με τον ε, Υπουργό των, τον ε, Επίτροπο για τι Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες εάν βρεθούμε μπροστά σε συνθήκες ισοδύναμες με αυτές τις πολύ δύσκολε που περάσαμε τα τελευταία χρόνια αλλά θα είναι σπανίο το πιστεύω να κληθεί ο πολίτης να πληρώσει επανειλημμένος για να διασώσει τράπεζες οι οποίες σε πολύ κρίσιμες χρονικές περιόδους ανέλαβαν υψηλότερα τους κινδύνους. Αυτό λοιπόν το θέμα των κρατικών ενισχύσεων ελπίζω ότι θα αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα πνεύμα της οδηγίας αυτής όπου θα ε, υπάρχει η διαδικασία του Μπέιλιν πρώτα πριν να χορηγηθούν οι εθνικές ενισχύσεις. Ευχαριστώ κυρία Σουίνμπορν από τους τηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία υποψήφια ο Πρωθυπουργός και Υπουργό των και ο Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου έκαναν μία πρόταση για αυτό που ονομάζεται διπλή, διπλό Ιρλανδικό παιχνίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο για ε, διάσωση. Ωστόσο υπάρχουν πολλές ε, κατηγορίες εις βάρος της Ιρλανδικής κυβέρνησης για την ε, φορολογική αντιμετώπιση επιχειρήσεων μεγάλων όπως τη Apple η οποία πληρώνει πάρα πολύ χαμηλούς φόρους. Ο Επίτροπος Αλμούνια ενημέρωσε τους Ιρλανδούς ότι οι ε, κανόνες, οι νόμοι που είχαν εγκρίνει το 2001 και το 2007 ήταν ε, ε, παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού και ως εκ τούτου θα υπάρξουν συνέπειες. Ερωτώ λοιπόν, εάν αγοράζονται σε ένα κομπιούτερ εγώ αυτή τη στιγμή της Apple, παραβιάζω το δίκαιο περί ανταγωνισμού και επίσης τι είδου πρωτότυπα μέσα μπορεί να βρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αντιμετωπίσει κανόνες οι οποίοι ε, παραβιάζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Ένα από τα, τα που διδάχθηκα αυτή την εβδομάδα είναι ότι διπλός Ιρλανδικός δεν σημαίνει καφές. Είναι μια πολύ ε, ζωφερή ρύθμιση. Πολλά είναι τα ε, πολλές είναι οι ερμηνείες του Double Irish σε διάφορους όρους της αργό που θα προτιμήσω να αποφύγω για να μην μπούμε σε ολιστερά πεδία. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι το εξή ότι οι εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλουν τον εταιρικό φόρο. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ποιε είναι αυτέ οι μεγάλε εταιρείε οι οποίε μπορούν να βρουν ειδικέ ρυθμίσει ώστε. Τουλάχιστον αυτό υποψιαζόμαστε προς το παρόν, να ε, βρουν ευολικέ ε, βολικές φορολογικές υποστάσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να πληρώνουν χαμηλότερο φόρο. Το ξεκίνησε ο Επίτροπος Αρμούνια. Θα συνεχίσω εγώ τη διερεύνηση για να ρίξω πλήρες φως όσο γίνεται. Απολύτως σεβαστό είναι το γεγονός ότι τα θέματα της φορολογικής πολιτικής απαιτούν ομοφωνία δεν θα προσπαθήσω να βάλω από την πίσω πόρτα μια ενοποίηση της πολιτικής της φορολογικής. Αλλά εάν αυτό ισοδυναμεί άμεσα ή έμεσα με ενισχύσεις προφανώς αφορά και το χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ερευνούμε τα τεκτονόμενα, τα έσοδα, το τι μπορεί να ε, προξενηθεί ως πρόβλημα και πώς θα δώσουμε τέρμα στο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σιλβί Γκουλάχ εκ μέρους των, ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σημειώσω, κυρία μου, κυρία Βέσταγκερ, ότι λυπούμε πολύ που είναι τόσο λίγοι παριστάμενοι σε αυτήν εδώ την ακρόαση και όχι επειδή είμαι και εγώ φιλελεύθερη, αλλά γιατί είναι μάλλον η πιο σημαντική ακρόαση αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν βλέπω πώς είναι οι Γάλλοι ε, συνάδελφοι οι οποίοι ε, προξενούν προβλήματα σχέση με την πολιτική του ανταγωνισμού, καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερους παρόντες εδώ σήμερα. Λυπούμε πολύ λοιπόν. Ξεκινάω με αυτό. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι μέσων επιβολής της δικαιοσύνης είναι αυτό που επιτρέπει στον ε, νεοεισερχόμενο στον επιχειρηματικό κόσμο να έχει ισοδύναμες ευκαιρίες με τους πιο μεγάλους ε, και γι' αυτό εδώ πολύ σωστά τοποθετηθήκατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση. Αλλά εδώ και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπάλς, υπάρχουν, υπάρχει εντύπωση για ορισμένους πολίτες από αυτό που συμβαίνει σχέση με μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι, δικέ ότι οι δικές μας επιχειρήσεις που βρίσκονται απέναντι σε μεγάλες του διεθνούς ε, ανταγωνισμού, ε, εκτεθειμένες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ότι ο δικό, η δική μας κανόνα του ανταγωνισμού είναι αυτές, αυτοί που τις θέτουν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό. ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ πλήρως ότι αυτή μπορεί να είναι η εντύπωση που δημιουργείται γιατί την εντύπωση τη δημιουργεί κανεί από αυτά τα οποία βλέπει στα μέσα ενημέρωση, αυτά που ακούει από τον περίγυρό του, ότι οι επιχειρήσει μα βρίσκονται σε δοκιμασία στο παγκόσμιο στερέωμα. Το καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανησυχεί του πολίτε μα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα να πούμε ότι στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι σαφέ ότι ο ανταγωνισμό θα οδηγήσει σε καινοτομία και σε ανάπτυξη, επομένω και σε θέσεις απασχολήσεως. Το βραχυπρόθεσμο όμως κόστος μπορεί να υπάρχει πράγματι. Είναι απαραίτητο εδώ να σκεφτούμε ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επανακατάρτιση των εργαζομένων για να αλλάξουν τομείς και ό,τι γίνεται θα πρέπει πάντα να συνάδει ε, με την αρχή της διαφάνειας και να μπορούν όλοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν να γίνονται πράγματα πάνω από το κεφάλι τους χωρί να έχουν καμία απολύτως συμμετοχή. Θα πρέπει να ακούσουμε περισσότερο τις απόψεις των απλών ανθρώπων. Δεν είναι υγιές το να θέλουμε να προσπαθούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τον ανταγωνισμό που έχει ακριβώς το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν και από ό,τι κατάλαβα αυτό το οποίο ρωτάτε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να πω είναι το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια εξισορροπημένη προσέγγιση και να βλέπουμε το σύνολο της εικόνας και όχι μονάχα ένα τμήμα της εικόνας. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Τι θα πείτε όταν μια ξένη εταιρεία αγοράζει μια ευρωπαϊκή εταιρεία με κρατική βοήθεια από μια άλλη χώρα, από μια εξωτερική χώρα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα, δυστυχώς πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν πάρει τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις και αυτές. Τούτου λεχθέντος όμως είναι απαραίτητο να το αντιμετωπίσουμε ανοιχτά. Να το συζητήσουμε όταν έχουμε εμπορικέ συμφωνίες, όταν συζητάμε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Να το συζητήσουμε λοιπόν με τους εταίρους μας, με τις αρχές ανταγωνισμού σε άλλες χώρες, για να καταλάβουν και αυτοί ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλιώς μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου μπαίνουμε σε μια κατερχόμενη σπήρα η οποία μας οδηγεί όλο και περισσότερο σε ένα ολιστήρο έδαφος εθνικών επιδοτήσεων και αυτό θα είναι πάντα σε βάρος των καταναλωτών. Η Ρίνα Κάρη από την ΚΟΥΕ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εδώ Τι κάνει. Σας ευχαριστώ. Ε, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ε, όταν σαν παράδειγμα ένας δήμος κάνει μια μεγάλη επένδυση για να φτιάξει μια υποδομή σημαντική όπως ένα τμήμα μετρό ή κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα και μια ρήτρα η οποία δίνει την δυνατότητα να δανειστεί κάποια χρήματα ίσως αλλά η πρακτική αυτή δυσκολεύεται τελευταία σε σχέση με τους κανόνες, με το σεβασμό των κανόνων ε, για τον ανταγωνισμό. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε και στις ε, δημόσιες προμήθειες ή τις προμήθειες τις οποίες κάνουν οι τοπικές αρχές την δυνατότητα να μπορούν να λειτουργούν και στα πλαίσια των κανόνων που διέπουν και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εσείς ε, αναφερθήκατε ίσως σε δικαστικές αποφάσεις. Το πρόβλημα εδώ είναι και ο χρονισμός με τον οποίο εκδίδεται μία απόφαση και ε, ο τρόπος με τον οποίο καλείται να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό εδώ είναι να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και μέσω των ΣΤΑΖ στις ιδιωτικές και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Όταν υπάρχει σαν παράδειγμα ε, μια προκήρυξη ε, πρέπει να ε, υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες να καλύπτουν και την δυνατότητα οργάνωσης ΣΤΑΖ για την κατάρτιση του προσωπικού. Το θέμα είναι βέβαια όλοι να υπακούν στους ίδιους κανόνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο θα συζητήσουμε πολλές φορές στο μέλλον. Thank you. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Μάικλ Γάιμον. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές αναφέρατε στην εισαγωγική σας παρατήρηση ότι θέλετε να υποστηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό των μεγάλων. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δύο εβδομάδε πριν τη Δευτέρα, ο Επίτροπο Αλμούνια στην Επιτροπή μα, ε, αναφερόμενο σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο του Ηνωμένου Βασιλείου, μα είπε ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί η απόφαση για την ε, υπόθεση αυτή, γιατί πρόκειται για μια ενίσχυση με τη μορφή τιμή διπλάσια από αυτήν τη αγορά και ω εκ τούτου ε, δυσμενείς συνθήκες ανταγωνισμού για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ρωτήσω εσάς, όταν πρόκειται να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα για την νέα Επιτροπή, τι θα πρέπει να περιμένουμε, τι θα πρέπει να γίνει σε αυτή την υπόθεση του πυρηνικού, των πυρηνικού εργοστασίου, πώς θα πρέπει να εξελιχθεί, τι είδους στάση και αντίδραση θα έχετε ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί ε, ανάλογα με την απόφαση του κυρίου Αλμούνια. Το έχει υπογράψει ο κύριος Αλμούνια. Θα συνεχίσετε. Εφόσον έχει ληφθεί η απόφαση, δεν νομίζω ότι θα έχω εγώ να κάνω κάτι, λέει η κυρία Βεστάγκερ από ό,τι βλέπω έχει τύχει επεξεργασίας και προετοιμασίας όλη αυτή η υπόθεση επί διετία. Εάν θεωρεί ο Επίτροπος ότι είναι όριμη η υπόθεση για να υποβληθεί στην ε, Επιτροπή ως λογικό όργανο, προφανώς δεν είναι έτσι. Αλλά να το πω διαφορετικά. Εάν προκύψει ισοδύναμη περίπτωση με αντίστοιχες περιστάσεις Σημαντικό είναι να γίνεται σεβαστό το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν μόνα τους το μείγμα ενέργειας ε, που θέλουν στην προμήθεια ενέργειας και στην παραγωγή ενέργειας. Δεν είναι δικό μας καθήκον, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και άρα, ως προς αυτό, σημαντικό θα είναι να ε, τηρούνται οι κανόνες του ανταγωνισμού. Οι κανόνες περί κρατικών ανησύσεων να μην υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα ή τέλη, οτιδήποτε γίνεται να γίνεται σε ισότιμους όρους και χωρίς ε, έμεσες ε, ή κρυφές κρατικές ενισχύσεις. Αυτό ήταν ε, μέχρι τώρα από ό,τι κατάλαβα το καθήκον του Επιτρόπου και του προσωπικού του, να διερευνούν δηλαδή τέτοιου είδους υποθέσεις και αυτή θα είναι και η βάση πάνω στην οποία ληφθεί η απόφαση ή θα ληφθεί η απόφαση. Ο καθένας μπορεί να έχει την δική του γνώμη να είναι υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, δεν κρίνεται αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αποφασίζουν τα κράτη-μέλη προς προ το μείγμα ενέργεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει απλώ να εξασφαλίζει ότι εάν ε, τίθεται ζήτημα κρατικών ενισχύσεων, αυτέ θα είναι συμβατέ με τη συνθήκη. Ευχαριστώ. Για την ομάδα EFTD ο Στέφεν Γούλφ. Καλησπέρα σας κυρία Βέσταγκερ. Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο μπήκε το 1973 στην κοινή αγορά. Εμείς θεωρούσαμε ότι θα μπαίναμε σε μια ευμαρή οικονομική ένωση. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου 40% της παγκόσμιας παραγωγής. Από τότε που αποφασίστηκε να γίνει μια πολιτική ένωση, σαν ένα κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πια μόνο 25% του παγκοσμίου εμπορίου και σε 10 χρόνια θα έχει πέσει στα 15%. Λόγω των υψηλών φορολογιών, της υπερβολικής ρύθμισης και που οι ανταγωνιστές μας, όπως και η κοινοπολιτεία που έχουμε αφήσει πίσω όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα είναι σε καλύτερη θέση από εμά. Όλα αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρόνια. Μήπως θα συμφωνούσατε ότι δείχνουν τα στοιχεία ότι δεν βοήθησε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταγωνιστούν εναντίον μηδενός. Με κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζω αυτή την εικόνα που μου παρουσιάζεται της Ευρώπης ως την Ευρώπη που πιστεύω εγώ σε αυτήν, ούτε για το παρελθόν, ούτε για το μέλλον. Κάθε άλλο. Αυτό που το οποίο έχω δει είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει αναπτυχθεί από μια κοινή αγορά μονάχα σε μια κοινότητα αλληλεγγύης και αλληλοεξάρτησης και όπου υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και αυτού που κάνουμε από κοινού. Και νομίζω ότι η ευμάρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητα να αντιμετωπίσει και να συγκρατήσει, τα αποτελέσματα μιας μεγάλης κρίσης όπως αυτή που περάσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους μη εγγεγραμμένους ο Σωτήριος Αριανόπουλος. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, επιτρέψτε μου μία επισήμωση διαδικαστικό ζήτημα. Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν αποτελούν πολιτική ομάδα, δεν έχουν νέο εκπρόσωπο, οπότε δεν τους εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ μόνο το κόμμα με το οποίο κλαίθηκα στη χώρα μου. Τώρα επί του θέματος. Ε, κυρία υποψήφιε, στο όνομα της, ε, του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε αυτή και εσείς βεβαίως με τη σειρά σας μείωση τιμών και νέες θέσεις εργασίας αλλά αντί αυτόν είδαμε μεγαλύτερη συγκέντρωση δύναμης στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, υψηλότερες τιμές έκρηξη της ανεργίας και μείωση μισθών. Στη χώρα μου στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες τα πάντα ιδιωτικοποιούνται. Αεροδρόμια, λιμάνια, ενέργεια, το νερό το ίδιο. Παραδίδονται σε μεγάλους ομίλους που απολύουν εργαζόμενους και αυξάνουν τις τιμές. Κρατικές παραγωγικές δομές, για παράδειγμα η αμυντική βιομηχανία, απαξιώνονται και παραδίδονται σε μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους. Η ελευθερία κίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων κυριολεκτικά διέλυσε κλάδου, έκλεισε επιχειρήσει γιατί βρήκαν ευθυνότερε αγορές εργασίας αλλού και απολύθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Οι τράπεζες συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται με πακτολό χρημάτων για να ε, ικανοποιήσουν υγιείς επιχειρήσεις, δηλαδή μεγάλες. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, γιατί είχατε το διαδικαστικό ζήτημα. Δηλαδή θα πάρουν πάλι κεφάλι έναντι των μικρών επιχειρήσεων. Ποιον τελικά ωφελούν αυτά. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, δείχνετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου να απαντήσω σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να αναγνωρίσουμε ότι ανεξάρτητα με το βλέμμα που έχει κανείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενσυναίσθηση, η συμπόνια για τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτήν την οικονομική κρίση είναι κοινή σε όλους. Αυτό ισχύει και για τους νέους στην Ελλάδα και για τους νέους στην Πορτογαλία και για τους νέους στην Ισπανία που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, που δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια πορεία, μια σταδιοδρομία, δεν μπορούν να αρχίσουν μια οικογένεια γιατί δεν έχουν τρόπο να τη Αυτό ανεξαρτήτως κόμματος και ανεξαρτήτως της θεώρησης που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το, το, συναισθανόμαστε όλοι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αναγνωρίσω ή να δεχθώ ότι είναι υπέτεια γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παράγων σοβαρότατος της λύσης. Γιατί ο, η παγκοσμιοποίηση είναι όλο και μεγαλύτερη και άρα οι χώρες μας γίνονται όλο και πιο μικρές και όλο και πιο αλληλεξαρτώμενες η μία από την άλλη. Και γι' αυτό εγώ στηρίζω αυτή την υπόσχεση σε μια ευκαιρία συνεργασίας μαζί σας γιατί το βρίσκω πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το να δείξουμε ενσυναίσθηση και συμπόνια στους ανθρώπους αυτούς που υποφέρουν πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός μιας συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου για να χτίσουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Μια ισχυρή Ευρώπη που δεν χτίζεται όταν την κατηγορούμε για οποιοδήποτε δεινό έχει συμβεί, ανεξαρτήτως της προέλευσης και της καταγωγής μας. Ευχαριστώ πολύ. Λουδεκνίδε Μάια. Γεια σας. Εγώ εξετίμησα δεόντως και τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα και την εισαγωγική σας παρέμβαση. Αν είστε τόσο επακριβείς και αυστηροί με το χρόνο σας στη δουλειά σας όταν την ξεκινήσετε όπως ήσασταν στην εισαγωγική σας παρέμβαση όλα θα πάνε καλύτερα στην Ευρώπη. Εγώ συμμερίζομαι τις αξίες τις οποίες αναφέρατε για την Ευρώπη, πρέπει όμως να πούμε ότι μερικές φορές ε, υπερβάλλουμε σε επίπεδο διακανονισμών και νόμων και κανόνων. Η ανησυχία μου είναι ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις μερικές φορές βασίζονται στη λογική κτλ. Δεν λειτουργούν όμως πάντα με τον θετικό τρόπο που θα έπρεπε. Παρακαλώ τι μπορείτε να κάνετε ως Επίτροπος έτσι ώστε να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις μόνο εάν αποδεικνύεται ότι τα ωφέλη είναι περισσότερα του κόστους και εφόσον πάντα όλα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν σε ένα κλίμα βελτιωμένης διαφάνειας. Θα συμφωνήσω ότι οι κανονισμοί και οι νομικές ρυθμίσεις δεν είναι πάντα ο σωστός ο δρόμος και το λέω αυτό γιατί αλλιώς δεν θα ήταν εύκολο να είμαι ε, επίτροπος για τον ανταγωνισμό. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν νέες ιδιαίτερα πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις. Η διαφάνεια λοιπόν, η σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, οι νέοι τρόποι συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν δρόμοι τους οποίους πρέπει να ανοιχνεύσουμε. Αυτό το οποίο όμως θεωρεί σημαντικό, θεωρώ σημαντικό για να μπορέσω λίγο να έχω μια ισορροπημένη άποψη είναι ότι στην ουσία ο ευρωπαϊκός τρόπος ρύθμισης ε, και διακανονισμού αντικαθιστά άλλους 28 αυτό είναι ένα πρόβλημα η, ρύθμιση αυτή βέβαια, αλλά εξυπηρετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σαν παράδειγμα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν ε, τι σημαίνει και τι συμβαίνει σε κάθε χώρα σε επίπεδο ε, ρυθμίσεων και νόμων. Ε, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στις ε, διάφορες αγορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές να κατανοήσουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές. Σαν παράδειγμα τα τραπεζικά τέλη στις πληρωμές. Υπάρχουν κρυφά τραπεζικά τέλη μερικές φορές. Εκεί υπάρχει μια αδυναμία γιατί σαν πελάτες δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτήν την διαδικασία και ίσως εκεί να χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Αλλά πάντως εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να προωθήσω μια ισορροπία ανάμεσα στην νομοθετική ρύθμιση από τη μία και στη χρήση άλλων μέσων από την άλλη έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Σας ευχαριστώ. Η Ανελίζε Ντόντς. Να σας συγχαρώ και εγώ για την ε, πρόταση διορισμού σας. Ε, υπάρχει ευκαιρία μεγάλη ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν σε αγορές οι οποίες κυριαρχούνται από τεράστιες επιχειρήσεις. Σαν παράδειγμα αναφέρομαι σε κάτι που γνωρίζω καλά, η ενέργεια ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχείται από έξι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν κάποτε περιφερειακά μικρά μονοπόλια και ε, από κοινού καλύπτουν το 95% της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και, γνωρί, και κατέχουν το 80% άνω το 70% εν πάση περιπτώσει της παραγωγής ενέργειας. Ε, αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο πληρώνουμε πάνω από 160-170 ευρώ κάθε οικογένεια επιπλέον γιατί ακριβώς δεν ε, λειτουργεί σωστά η αγορά. Να λοιπόν ένα παράδειγμα ενός προβλήματος το οποίο δεν ισχύει μόνο στη χώρα μου αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μικρές επιχειρήσεις αποκλείονται από τις αγορές εις βάρος ε, των πολιτών των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε σαν επίτροπος για να αντιμετωπίσετε αυτού του είδους τα θέματα. Well, ευχαριστώ για το αυτό. Για το συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα, γιατί αυτό δείχνει τι αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Ότι η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί όπως θέλουμε να λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχει Πραγματικό ανταγωνισμό, υπάρχουν μερικέ κυρίαρχες εταιρείε που έχουν μοιράσει την αγορά μεταξύ του και είναι πολύ δύσκολο για του καταναλωτέ να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή του ω καταναλωτές για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία που έχω στα χέρια μου για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι οι κανόνες που έχουν να κάνουν με τη νομοθεσία antitrust και κατά τον... Ε, ε, συγχωνεύσεων και για να επαλέφθω σε αυτό που είπατε για τον πυρικό σταθμό του Χίνκλεϊ, οι κρατικές επιδοτήσεις. Και παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι ερωτευμένη με τον ανταγωνισμό, πάντα γίνεται έτσι. Στην αρχή, τουλάχιστον, υπάρχουν όρια ακόμα και σε αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό προσβλέπω στη δυνατότητα να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν για τα θέματα αυτά, με τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση και με τον Επίτροπο, ο οποίος ε, ασχολείται με τα θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, γιατί με τα διαφορετικά αυτά εργαλεία μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Έχω ακούσει κάτι αριθμητικά ποσά που είναι τεράστια για το πόσο πρέπει να επενδύσουμε για να έχουμε την ενεργειακή υποδομή που θέλουμε τα επόμενα 15 χρόνια. Νομίζω ότι να, το να εργαστούμε από κοινού για αυτά τα προβλήματα και το να εφαρμόσουμε τους κανόνες που έχουμε στη διάθεσή μας θα βοηθήσει τους καταναλωτές να έχουν μικρότερο τιμήμα για την ενέργεια. Από την Επιτροπή ΙΜΚΟ ο Ανδρέας Σφάμπ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποψήφια Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα περίπλοκα ζητήματα είναι πολύ σαφής και απλή και νομίζω ότι είναι κατανοητή και για τον κάθε πολίτη, για το τι σημαίνει ανταγωνισμός. Θα ήθελα λοιπόν να μπω σε ένα κάπως περίπλοκο ζήτημα. Γι' αυτό ξεκινάω λέγοντας εν γέννη ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που δίνεται έμφαση στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Όμως το ζήτημα του ανταγωνισμού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εναντί των μεγάλων, ε, διότι ο κύριος ε, κανονισμός θεωρεί ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις το 10% του ε, καρτέλ όταν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις ε, το προϊόντος καρτέλ δηλαδή 10% ενώ οι μικρότερες, έχουν, μικρότερες επιχειρήσεις έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο σαφή ρύθμιση ώστε οι κυρώσεις, το 10% δηλαδή από το προϊόν του καρτέλ, να μην είναι τόσο βαριές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, το καλύτερο είναι μην ξεκινάει κανείς να φτιάχνει καρτέλ, έτσι. Αυτό το λέω σαν συμβουλή για όσους μας ακούνε, όχι σας φυσικά. Και βεβαίως υπάρχει ζήτημα. Όταν έχουμε εταιρείε με πληθώρα χαρτοφυλακίων προϊόντων, φάσμα προϊόντων μεγάλο και άλλες επιχειρήσεις που έχουν ένα-δύο μόνο προϊόντα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Από τις υποθέσεις που μελέτησα μέχρι τώρα, διαπιστώνω ότι οι ρυθμίσεις που έχουμε, οι κανόνες που έχουμε για τα πρόστιμα, εξασφαλίζουν μια κάποια ασφάλεια δικαίου, με την έννοια ότι κανείς γνωρίζει ότι αν τον πιάσουν θα συμβεί αυτό και αυτό, από την άλλη, υπάρχουν και διατάξεις που επιτρέπουν να ληφθούν υπόψη ειδικέ περιστάσεις. Τι ρόλο έχει κανείς μέσα στο καρτέλ. Ήταν αυτός που το σχεδίασε, ήταν κάποιος που ακολούθησε, που θα έπρεπε να έχει πει μεν όχι, αλλά τελικά παρασύρθηκε και μπήκε μέσα. Άρα υπάρχει ένα ζήγισμα, μια στάθμιση της κατάστασης. Από την άλλη βέβαια, αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόστιμο να είναι αποτρεπτικό στο μέγεθός του. Διαφορετικά βάζουν ακόμα μια γραμμή στον ισολογισμό. Αντί να έχουν μεγαλύτερο κέρδος, ε, βάζουν και το πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσουμε. Δεν αρκεί αυτό όμως. Το πρόστιμο πρέπει να είναι τέτοιο και τόσο βαρύ ώστε να είναι αποτρεπτικό. Και όταν κανείς ενημερώνεται ότι μια άλλη επιχείρηση έχει φτιάξει καρτέλ, να λέει «Α, αυτοί με κοροϊδέψανε, με εξαπατήσανε, με ρίξανε» και άρα είναι η σειρά του τώρα να υποστούν τις συνθήκες, τις επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι η ε, επιπτώσεις, η κύρωση, το πρόστιμο τόσο υψηλό ώστε να μην αφήνει καμία ευκαιρία να φτιαχτεί καρτέλ. Ευχαριστώ Γέπε Κόφωτ, Σοσιαλιστές Δημοκρατές. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τη Μαργαρέτα Βέστεκερ για την πολύ ωραία ενακτήρια της ομιλία. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να είναι ένας πραγματικός πολιτικός και ένας πεπισμένος πολιτικός ο οποίος αντιμετωπίζει την πολιτική ανταγωνισμού και να αντιμετωπίσει και τους μεγάλους και τους μικρούς και να μπορέσει να προωθήσει την ανάπτυξη. Στην ε, επιστολή που αφορά την αποστολή σας που σας έδωσε ο κύριος Γιούγκερ αναφέρεται σαφώς ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ε, φοροαποφυγής που κάνουν διάφορες εταιρείες με την αρρωγή μερικές φορές ορισμένων κρατών μελών. Θα ήθελα να ξέρω όμως πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα, ώστε να μην μείνουν στο δινεκές αυτές οι υποθέσεις και να υπάρξει κάποια κύρωση και εναντίον των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες, γιατί αλλιώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τις εταιρείες να παίξουν με τα φορολογικά συστήματα. Ευχαριστώ για τα θερμά σου λόγια. σε σχέση με τα θέματα αυτά πρέπει να είμαι κατηγορηματική. Αν δεν έχουμε σαφείς κανόνες και σαφή αντιμετώπιση μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτό είναι μονάχα ένα τεχνικό θέμα. Δεν είναι καθόλου τεχνικό θέμα, είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Γιατί κάθε επιχείρηση θέλει να διερευνήσει νέες αγορές, θέλει να επενδύσει, να βρει καινούργιες αγορές. Οι μεγάλες εταιρείες όμως που έχουν τεράστια κέρδη και τεράστιους πόρους, αν τα καταφέρουν έτσι ώστε να πληρώνουν ένα πολύ μικρότερο ποσοστό των κερδών τους ως φόρους από τις μικρές επιχειρήσεις, τότε ουσιαστικά οι μικρές επιχειρήσεις πληρώνουν τους φόρους των μεγάλων. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η έρευνα η οποία πρέπει να γίνει να είναι πλήρης ώστε οι υποψίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν να διαλύονται. Υπάρχουν πολλές υποψίες, το θέμα είναι να μπορούμε να εξακριβώσουμε αν αυτές οι υποψίες ευσταθούν ή όχι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για τις έρευνες που είναι εν εξελίξη, αλλά θα ήθελα να μπορέσει να γίνει αυτό σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα προτεραιότητας, είναι ένα θέμα το οποίο είναι κέριο για τον ανταγωνισμό και εάν καθυστερούμε θα δώσουμε ένα πολύ αρνητικό συνιάλο για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ντάριος Ροζάτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου δεν είναι ισοδίκαια ούτε ανταγωνιστική. Υπάρχουν εξωτερικοί πάροχοι φυσικού αερίου που έχουν χρησιμοποιήσει τη δεσπόζουσα θέση του και έχουν εφαρμόσει διακριτικές πρακτικές έναντι των καταναλωτών. Μία από αυτές τις εταιρείες, η Gazprom, είναι διαβόητη για το ότι έχει εμποδίσει τη διαφοροποίηση των ε, προμηθειών φυσικού αερίου και εφαρμόσει πρακτικές αθέμη του ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, πολλές πολλοί καταναλωτές στην Ευρώπη πληρώνουν 78% περισσότερο ακριβό το φυσικό αέριο από ότι άλλους καταναλωτές. Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει μια ισοδίκια και ανταγωνιστική αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ξεκινώντας, οφείλω να αναγνωρίσω κάποια από τα μηνύματα τα οποία μας δίδεται σήμερα ότι κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτες ελέγχουν την αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι έρευνες για τις πρακτικές της εμπορικές της Gazprom θα συνεχιστούν. Δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, αλλά πάντως συνεχίζονται και κάποια στιγμή θα καταλήξουν. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εντάσσεται και στις προτεραιότητες του υποψηφίου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα λοιπόν, γιατί οι τιμές της ενέργειας είναι ο καθοριστικός παράγων για τη λειτουργία όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Συνεπώς, έχει σημασία να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τις έρευνες οι οποίες γίνονται και να βεβαιωθούμε ότι θα βελτιωθούν και θα εφαρμοστούν πλήρως όλοι οι κανόνες εναντίον των τραστ. Γιατί αν γίνει αυτό ίσως να δούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης και αν δεν το κάνουμε αυτό θα θελήσουν και άλλες επιχειρήσεις ε, να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πρακτικές και να δυσκολέψουν τις αγορές. Είναι σημαντικό θέμα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά γενικότερα για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, Άντερ Σπριμνταλ Βίστισεν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σήμερα αλλά και πιο παλιά έχετε τονίσει ότι λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις και επιλογές στον τομέα αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι θέλουν να αφήσουν καλύτερα κατά μέρο τις φιλελεύθερες αυτές επιλογές και να αφήσουν ένα περιθώριο για την ανάπτυξη νέων ε, κλάδων στην Ευρώπη. Έχουμε πρωταθλητές δηλαδή στην Ευρώπη στο πρόσωπο ορισμένων εταιριών. Εσύ όμω, ποια είναι η άποψή σου για αυτό το θέμα, πώ θα διαχειριστεί αυτή την τάση να αναδεικνύονται σε πρωταθλητέ ορισμένε επιχειρήσει και για αυτό το λόγο να χαλαρώνουν κάπω οι αγώνε, οι κανόνε ανταγωνισμού για να μπορέσουν να προκύψουν νέοι πρωταθλητέ σε βιομηχανικό επίπεδο στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξιών από το να έχουμε απλώς Ευρωπαίους πρωταθλητές. Πρέπει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι πρωτοπόρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επαναλαμβάνω. Μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί καλύτερα στις παγκόσμιες αγορές όταν μπορεί να ανταγωνίζεται στο δικό του χώρο. Και αυτό είναι απόλυτα σχετικό με αυτό που λες. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχουμε απλώς πρωταθλητές, κάποιος άλλος θα πληρώνει την ύφη. Αν περιορίσουμε τον ανταγωνισμό, τελικά ο κίνδυνος είναι ότι τα προϊόντα μας θα είναι πιο ακριβά και θα σταματήσουμε να καινοτομούμε και τελικά για τους καταναλωτές θα υπάρχουν πιο ακριβά προϊόντα τα οποία θα είναι χαμηλότερες ποιότητες. Αυτό πρέπει να πούμε σε αυτού που προτείνουν κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια δημιουργήση προταλυτών δεν είναι δωρεάν. Κάποιο πληρώνει το κόστο τη. Γι' αυτό για μένα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε όταν επιμένουμε ότι πρέπει να είναι χωρίς περιορισμούς η πολιτική ανταγωνισμού, τονίζω πάντα ότι για να μπορεί κανείς να είναι έξω ανταγωνιστικός πρέπει να είναι και μέσα στο ίδιο το σπίτι ανταγωνιστικός. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες που μπορούν ενδεχομένως να ευνοήσουν ορισμένε μορφές συνεργασίας όπως είναι οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και να μας ενισχύσει για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ρέμον Τρεμόσε Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Φεστάγερ, εάν προφέρω σωστά το όνομά σας, υποψήφια επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη νέα πνοή μετά τις ακροάσεις που έχουμε δει. Έκανα μια μικρή αναζήτηση στο Google για υποθέσεις αντιτράστ και ιδιαίτερα ήθελα να πω ότι εκτιμώ την αναφορά σας στον ψηφιακό χώρο, γιατί ξέρετε ότι η Google έχει ένα τεράστιο ποσοστό των, ε, των υπηρεσιών έρευνας στο ίντερνετ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει τρεις φορές την ευκαιρία στην Google να ε, κάνει διορθώσει έτσι ώστε να ε, σταματήσει την προτιμησιακή μεταχείριση των δικών της προϊόντων ως χρήση μηχανής αναζήτησης. Ε, ωστόσο αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει λύσει το ε, πρόβλημα, ούτε το να ανα, ανεβάσει στη σελίδα πιο πιο υψηλή θέση ανταγωνιστικά προϊόντα. Ε, ούτε είναι καν η καλύτερη λύση πάντοτε η αναζήτηση της Google ή τα προϊόντα της Google για τις, ως προς τις τιμές τους ή την ποιότητά τους. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κάτι. Η επιστολή ενστάσεων είναι το επόμενο βήμα για να προστατέψουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές μας. Απάντηση. αυτή την ώρα που μιλάω, δεν ξέρω ποιο είναι το συγκεκριμένο επόμενο βήμα. Αλλά επόμενα βήματα θα υπάρξουν, είμαι βέβαιη. Διότι έχουμε, να κάνουμε με μια κλασική περίπτωση. Έχουμε μια επιχείρηση με τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο μερίδιο αγορά. Έχουμε ε, διαμαρτυρίες από διαφόρους ανταγωνιστέ και διαφημιστέ. Εχθές ακόμη, αν δεν κάνω λάθο προέκυψαν νέα στοιχεία που εντάχθησαν στον δημόσιο διάλογο στη Γερμανία και δίνουν και νέες διαστάσεις για το πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των θεμάτων από την Google και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να μην συζητήσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα σήμερα αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι και τα μέσα θα έχουμε στη θέσή μας και τη βούληση για να διερευνήσουμε όταν έρθει η ώρα και τους νέους αυτούς τομείς που φαίνεται να ανοίγουν. Όπως είπα σε αγωγικές μου παρατηρήσεις, οι κανόνες περί ε, ε, είναι παλιοί όσο και η συνθήκη. Πολύ καλό αυτό. Αλλά για να τους εφαρμόζουμε σωστά πρέπει να είμαστε στην αιχμή όπως και οι νέες εταιρείε που μπαίνουν στην αγορά. Και αυτό είναι το δύσκολο. Γι' αυτό και ελπίζω ειλικρινά ότι δεν θα χρειαστεί να κρατήσει η έρευνα αυτή περισσότερο από ό,τι χρειάζεται και να παραταθεί ε, γιατί θα εναλλάσσεται με μια επιπλέον έρευνα κτλ. Γιατί αυτό είναι εις βάρος και του καταναλωτή και της επιχείρησης που χρειάζονται ανοιχτές αγορές και υπηρεσίες ποιότητας διαθέσιμα στον καταναλωτή. Επόμενα βήματα λοιπόν θα υπάρξουν. Τι είδους προσεχή βήματα όμως είναι πολύ νωρίς να σας το πω. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Φερνάντε από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλώ ήρθατε. Ο Γιούνκερ στην ομιλία του τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο είπε ότι η εσωτερική αγορά δεν έχει αυτομάτως προτεραιότητα και ότι οι κοινωνικοί παράγοντε θα πρέπει και αυτοί να δραματίζουν το ρόλο του στην Ευρώπη. Στα ισπανικά. Στην εκλογική μου το Μάιο ε, βρέθηκα στο Σαν Μαρτίν Αουρέλιο, σε ένα χωριό, μαζί με γονείς ε, και παιδιών που είχαν πνευματικές ε, αναπηρίες. Είχαν αγωνιστεί για πάρα πολύ καιρό για να μπορέσει η περιφερειακή κυβέρνηση να τους δώσει κάποιο κτίριο όπου να ζουν αυτά τα παιδιά και τα τελευταία χρόνια αυτή η Ένωση φρόντιζε με επαγγελματίε αυτό το, αυτό το νίκο. Αλλά με μια λανθασμένη εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού υπάρχει πίεση τώρα αυτές οι, οι υπηρεσίες να δίνονται οι υποστηρίξεις, οι επιδοτήσεις να δίνονται για ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί αυτό το, αυτός ο οίκος για παιδιά με πνευματικές αναπηρίες να περάσει στα χέρια μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Πώς θέλει ο κύριος Γιούνκερ, πώς θέλετε κι εσείς να εξασφαλίσετε την ισορροπία μεταξύ του ανταγωνισμού από τη μια μεριά και της διατήρησης του κοινωνικού αυτού τομέα, του φιλανθρωπικού τομέα που εκφράζει το ευρωπαϊκό ε, πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης και είναι και μια ελπίδα για τις οικογένειες που έχουν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα. Καταρχάς, αυτό το οποίο θα πρέπει να σεβαστώ είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν ισχυρές ευθύνες στο συγκεκριμένο τομέα. αυτό που ονομάζουμε εμείς ε, στα πλαίσια του ανταγωνισμού υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος ή καθολικού συμφέροντος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να, να το ορίσουμε καλύτερα. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες τις οποίες έχουμε. Σαν παράδειγμα φέρατε το θέμα της προστασίας και της φροντίδας αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο πάει στις αγορές, υπάρχει όμως και ένα κομμάτι το οποίο δεν πρέπει να πάει στις αγορές. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το ορίσουμε σε επίπεδο πολιτικό. Αν ένα κράτος μέλος θέλει πράγματι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα ελέγχονται στη χώρα τη συγκεκριμένη, αυτό θα πρέπει να το κάνει αφού ορίσει το ποιες είναι οι κοινωνικές ανάγκες, οι πραγματικές τις οποίες έχει. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή ε, κοινωνία στην οποία ζούμε να οριστούν σωστά αυτά τα πράγματα. Η πολιτική σε εθνικό επίπεδο είναι σε μόνιμο διάλογο με τους εκλογείς τους και ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο χρειάζονται και με ποιο τρόπο ε, το χρειάζονται. Ελπίζω οι οικογένειες αυτές να βρουν κάποια λύση γιατί πράγματι οι εποχές είναι πολύ σκληρές στη χώρα σας. Ευχαριστώ Βέρνερ Λάγκεν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέσταγκερ. Είσαστε ιδεώδης υποψήφια. Προέρχεστε από ένα κράτος μικρό, χωρίς διαφθορά. Ε, έχετε καθαρό μητρό, έχετε σπουδές καλές φιλελεύθερη. Ε, νομίζω ότι τα βάρη του παρελθόντος τα έχετε μπροστά σας, γιατί ο κύριος Αλμούνια δεν μπόρεσε να λύσει το θέμα του Google. Έχετε ακόμη το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σοβαρά μέτρα ε, για το φορολογικό dumping ακόμη ε, ενισχύει, ενώ η Δανία έχει υψηλό φορολογικό συντελεστή. Και από την άλλη έχει τεράστια εξουσία να επιβάλλεται ε, κυρώσεις πρόστιμα χωρίς να υπάρχει σε δημοκρατικό έλεγχο. Θέλω λοιπόν το εξή να ρωτήσω. Πώς σκοπεύετε στο μέλλον να αναπτύσσετε τις κατευθυντήριε γραμμές σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και όχι παρά το Κοινοβούλιο. Και αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη, θα χρειαστεί να εξηγήσουμε για άλλη μια φορά και να καταστήσουμε σαφή στην κοινή γνώμη τη σημασία του δικαίου του ανταγωνισμού. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση, πώς θα το κάνετε δηλαδή. Τρίτη ερώτηση, πώς νομίζετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο στην προσεχή ε, περίοδο. Απάντηση. Καταρχάς, ελπίζω να είσαστε έτοιμος να πιείτε πολλούς καφέδες μαζί μου. Γιατί δεν Δανία έτσι τα λύνουν τα προβλήματα. Μια και δεν μπορούμε να καπνίζουμε πια, τώρα πίνουμε καφέδες. Και έτσι ξεκινάει ένας καλός διάλογος. Βέβαια, το θέμα του ανταγωνισμού είναι πολύ ειδική περίπτωση. Γιατί με το άρθρο 103 της συνθήκης έχουμε πολύ περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης ε, ε, έρευνας εποπτείας σε μια νομοθετική διαδικασία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης να γίνεται και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση με εσάς ε, όταν περνάμε σε ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν του υπείου δικαίου, του ενδοτικού δικαίου και να είμαστε σύμφωνοι πριν βάλουμε το μολύβι πάνω στο χαρτί και γράψουμε τη ρύθμιση. Η μέχρι τώρα στάση του Κοινοβουλίου ήταν πολύ χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη στήριξη στην εξέβρεση ε, της χρυσή τομή. Όπως είπα και νωρίτερα, θα πρέπει πάντα να κοιτάμε τη λογική εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη διαφάνεια, την ε, ρύθμιση της αγοράς, αλλά και για το θέμα που αναφέρεται. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να ξέρουμε ότι μπορεί να μην υπάρξει νομοθεσία, μπορεί να μην υπάρχει η συνήθις διαδικασία, αλλά μπορεί να υπάρχει έντονη επίδραση από πλευράς του Κοινοβουλίου και τήρηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των υποσχέσεών της είτε με τυπικό είτε με άτυπο τρόπο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη δεύτερη ερώτηση πρέπει να πω ότι δεν τη θυμάμαι, αλλά για την τρίτη ερώτηση. Α, πολιτική για την ενημέρωση προς τον καταναλωτή, προς τον ε, πολίτη. Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κινούμεθα, να έχουμε, ε, να απαντάμε ερωτήσεις, να έχουμε διαφάνεια όταν έρχονται αισθήματα στη Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, να είναι ανοιχτά αυτά που κάνει. Αλλά και για μένα πρέπει να είναι διαφανή στη στάση μου, να ξέρει ο κόσμος με ποιον συναντιέμαι, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε είναι κρατικές αρχές είτε είναι επιχειρήσεις. Η διαφάνεια είναι πάρα πολύ καλό μέσον στην υπόθεση αυτή. Και πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε μαζί στην επόμενη πενταετία, θα μπορέσουμε στο τέλος της πενταετίας να πούμε ότι τα καρτέλ τα φέραμε σε δύσκολη θέση. Θα μπορέσουμε να πούμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις ήταν, με υπεύθυνη στάση των κυβερνήσεων και ότι δώσαμε σαφή εικόνα και επισκόπηση στον πολίτη για το πώς χρησιμοποιήθηκε το χρήμα του και ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συμβάλει στη δημιουργία των θέσεων εργασία που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σίγουρα αυτό ε, ισχύει πάντα όταν ζητάμε αποζημιώσεις, όταν επιβάλλουμε πρόστιμα για αποζημιώσεις μέσα στη διαδικασία στην απόφαση. η Μαρίζα Ματίας τώρα για την ΚΟΕ. Εδώ είμαι κυρία υποψήφια επίτροπε ε, είστε η μόνη ουσιαστικά εκπρόσωπος από μια ριζοσπαστική αριστερά στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα. Μιλήσατε πάρα πολύ για την σημασία του ανταγωνισμού. Θα ήθελα απλώς να θέσω το ερώτημα αν θεωρείται ότι υπάρχουν και όρια στην πολιτική ανταγωνισμού. Αν θεωρείται ότι υπάρχουν κάποιοι τομεί που πρέπει να μείνουν έξω από το χώρο του ανταγωνισμού και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι τομεί. Μερικέ φορέ φοβάται ο κόσμο όταν ακούει μεταφρασμένο κατά λέξη ε, το όνομα του κομματός μου. Μιλάμε για ριζοσπαστική αριστερά, πρέπει να με προσέχετε. Αλλά σοβαρά τώρα, σε επίπεδο πολιτικό μας ονομάζουν και μας περιγράφουν σαν κοινωνικοφιλελεύθερους. Νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχουν όρια στον ανταγωνισμό, αυτό είναι σαφές. Και υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να, να δημιουργήσει ο ανταγωνισμός και γι' αυτό ακριβώς στην εισαγωγική μου παρέμβαση προσπάθησα να πω ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ένα μοναχικό χαρτοφυλάκιο. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι πρέπει να συνεργαστούμε σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών και σε επίπεδο επιτρόπων ε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, Εκτιμώ το όραμα του κυρίου Γιούνκερ για τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, θα εργαστούμε και ε, με τις προοπτικές για τους νέες θέσεις αντιπροέδρων. Ένα άλλο θέμα το οποίο με ικανοποιεί είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτό το οποίο από κοινού κάνουμε και σε αυτά τα οποία κάνουν τα κράτη-μέλη. Οι χώρες ε, είναι χώρες οι οποίες έχουν ε, τα κοινοβούλια των κρατών τους, ε, είναι σε στενή επαφή με τις εκλογικές τους περιφέρειες και γνωρίζουν τις πραγματικές τους ανάγκες και γι' αυτό ακριβώς εκτιμώ το ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ε, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό δεν θα το αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω τίποτα να πω εγώ σε αυτό αν μου επιβεβαιώσετε την επιλογή μου στη θέση του Επιτρόπου. Ευχαριστώ. Έρνες Τουρτασούν, ε, Πράσινη. Επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ισπανίας και των θεμάτων που αντιμετώπισε ο προκάτο ο κύριος ε, Αλμούνια. Το αποτέλεσμα είναι ότι, που έχει ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή οι, οι καταναλωτές στην Ισπανία πληρώνουν το πιο ακριβό ρεύμα, ενώ οι επιχειρήσει έχουν μια προνομιακή μεταχείριση. Έχουμε μια ολιγοπολιακή αγορά ενέργειας και αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση της οδηγίας 2072 που γνωρίζετε πολύ καλά για τους κοινούς κανόνες στον τομέα της ενέργειας. και πάρα πολλοί στην Ισπανία ζητούν ένα νέο υπόδειγμα για την ενεργεια, ενεργειακή πολιτική. Πώς θα προχωρήσετε για να υπάρχει η εφαρμογή αυτής της οδηγίας, να διαχωριστεί η εταιρεία που έχει την υποδομή και η εταιρεία που παράγει ηλεκτρισμό. Και πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει πραγματικά δυνατότητα ανταγωνισμού για τους μικρούς παραγωγούς στην Ισπανία που αυτή τη στιγμή είναι τελείως έξω από το κύκλωμα. I find this extremely Το θεωρώ ιδιαίτερα περίπλοκο αυτό όλο. Διότι αυτό που συνέβη την τελευταία διετία ήταν ότι κάποιες, κάποια κλάδη απο, απελευθερώθηκαν τελείως, ενώ κάποια άλλοι έμειναν όπως ήταν. Και προχωράμε με πολύ βραδείς ρυθμούς. Νομίζω ότι είναι η ώρα πια και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια ένωση ενεργειακή που θα μας δίνει με ασφάλεια, ενέργεια, σε οικονομικούς όρους ανεκτούς, φθηνή. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μια χώρα χωριστά. Για το θέμα βέβαια το πού χρειάζονται οι επενδύσεις, ασφαλώς η απάντηση είναι στον ενεργειακό τομέα και ως προς το δίκτυο διανομής και ως προς τους μηχανισμούς του δυναμικού ώστε να μπορούμε να ε, έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία στην ε, παραγωγή ενέργειας, αλλά τούτων λεχθέντων. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι επίτροποι και αντιπρόεδροι της Επιτροπής θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, νομίζω, εφόσον εγκριθώ στη θέση του Επιτρόπου της, ε, του ανταγωνισμού, να ερευνώ και αν κάποια επιχείρηση αξιοποιεί δεσπόζουσα θέση και άρα δυσκολεύει την είσοδο στην αγορά και την προμήθεια σε χαμηλότερη ε, τιμή για τον καταναλωτή ε, ενός μικρότερου ανταγωνιστή, ενός μικρότερης επιχείρησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα και επίσης μπορεί ένα τεράστιο βήμα μεν, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο και βήμα για να προχωρήσουμε, το να προχωρήσουμε σε μια ενεργειακή ένωση. Ευχαριστώ Τσάνι, η FTD. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησαν έρευνες για τις παραβιάσεις των κοινοτικών κανόνων για τον ανταγωνισμό από πλευράς της χώρας του Λουξεμβούργου και της εταιρείας Fiat. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού δηλαδή, είναι ένα απαράδεκτο σκάνδαλο. Ε, ποια είναι η γνώμη σας γύρω από αυτό και θα ήθελα να μάθω τον τρόπο με τον οποίο θα παραμβαίνετε για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό ε, με διαρθρωτικό τρόπο και εκ των προτέρων. Έχετε συζητήσει το θέμα Fiat με τον κύριο Γιούνκερ όταν ήταν ε, ε, πριν ένα χρόνο πρωθυπουργό του Μεγάλου Δουκάτου έλεγε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις φήμες για πιθανή έρευνα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, σωστότερη και διαρθρωτική αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Ένα πράγμα είναι το να ερευνά κατά περίπτωση ε, τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να είναι σαφή, σαφείς οι αρχές οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές θα πρέπει να πληρώνει κανείς τον φόρο που του αναλογεί, τον φόρο που του πληρώνουν οι ανταγωνιστές του, τον φόρο που πληρώνουν οι άλλες επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι το σωστό και δίκαιο. Όσο ε, σορεύουμε εμπειρίες μέσω των ερευνών αυτών, τις οποίες διεξάγουμε, Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε δύο πράγματα. Καταρχάς θα λειτουργήσουμε αποτρεπτικά και δεύτερον θα συλλέξουμε και πολλές γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτά τα, αυτές οι διαδικασίες. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ε, να μην εφαρμόζονται φορολογικές εθνικές πολιτικές από την πίσω πόρτα, γιατί τότε πράγματι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από ό,τι διαβάσαμε μέχρι τώρα, από τον τύπο τουλάχιστον, πράγματι πολλοί φαίνεται ότι θίγονται από αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί εκτιμούν όταν μία επιχείρηση πληρώνει σωστά τους φόρους της. Θα συνεχίσουμε τις έρευνες λοιπόν, οι οποίες όπως είπατε έχουν ξεκινήσει, θα προσπαθήσουμε να επωφεληθούμε από την εμπειρία που σωρεύουμε και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με πιο διαρθρωτικό τρόπο τα θέματα αυτά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το σύστημα προστασίας που εισάγει η οδηγία για τους δικαιούς όρους της καταναλωτικές συμβάσεις θεωρεί ότι βρίσκεται σε υποδέστερη έναντι του πολιτή ή προμηθευτή θέση ο καταναλωτής και ως προς την διαπραγματευτική του δύναμη και ως προς τις γνώσεις του. Αυτό που διαβάζω είναι ε, τμήμα μίας πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη ερμηνεία και εξήγηση αυτής της σχέσεως μεταξύ μιας τράπεζας και ενός δανειζομένου σε περίοδο οικονομικής κρίσεως και ιδίως στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ και προφανώς έχω υπόψη την πατρίδα μου την Κύπρο. Πιστεύετε ότι έχει έρθει η ώρα για μια πιο συγκεκριμένη πολιτική, για πιο αποφασιστική προστασία όλων αυτών των δανειστών από τις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές και πιστεύετε ότι έχει έρθει η στιγμή για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα δίνει την έμφαση στην ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας. Απάντηση. Ασφαλώς και το πιστεύω. Διότι τα τρία χρόνια αυτά που παρακολουθούσα τις συνεδριάσεις του ΕΚΟΦΗΝ, που ήμουν παρούσα στις συνεδριάσεις του ΕΚΟΦΗΝ, ακριβώς πάνω σε αυτό δουλεύαμε. Σε νέες και πιο αυστηρές απαιτήσει για αδίποτε ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Είτε είναι τράπεζα αυτό, είτε άλλος φορέας, άλλου τύπου ίδρυμα και ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσει και ως προς την ρευστότητα, την ε, στεναρότητα, την διακυβέρνηση έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν λήξει η κρίση θα έχουμε μια διαφορετική, ίσως και πιο βαρετή εικόνα του τραπεζικού τομέα. Και βεβαίως πρέπει να μεριμνήσουμε αυτοί οι κανόνες το όντι να εφαρμόζονται η Τραπεζική Ένωση θα προσφέρει πολλές από τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Η ενιαία εποπτεία θα λύσει κάποια άλλα προβλήματα. Επίσης θα υπάρξει και ζήτημα επιβολής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Διότι η Τραπεζική Ένωση δεν αποτελεί τη λύση απαραίτητα για τους πάντες και ότι είναι ανοιχτή και προς τις χώρες εκτός ευρώ. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα, οι, εισρωές και οι εκροές θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και αυτό σημαίνει και κρατικές ενισχύσεις. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό που έχει επεξεργαστεί το ΕΚΟΦΗΝ και με πολύ ισχυρή υποστήριξη και νομοθετική παρέμβαση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μία πρόταση που θα δώσει ισορροπημένες λύσεις εάν ξαναχρειαστεί να ε, αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ. Ζίκφριτ Μούρετσαν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τέθηκε το θέμα και από άλλους συναδέλφους ότι η πολιτική του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί προβλήματα ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, συνενώνονται κάποιες από αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές απορροφώνται από άλλες επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο δεν είναι ευνοϊκό για την παρουσία μας στην οικονομική στον κόσμο. Ε, πολλές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για αυτή την τάση. Ποια είναι η δική σας άποψη. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει την πράσινο φως για την συγχώνευση της Τελεφώνικα με την άλλη ισπανική επιχείρηση. Πιστεύετε ότι αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί την ανάγκη δημιουργίας μεγάλων παικτών στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό το οποίο έχει σημασία όταν μιλάμε για συγχωνεύσεις στις αγορές είναι να κατανοούμε καταρχάς το πώς λειτουργούν οι αγορές. Γιατί πράγματι πρέπει κάθε φορά να το βλέπουμε το πράγμα με ξεχωριστό τρόπο. Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο δηλαδή. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν οι συγχωνεύσεις να γίνονται δεκτές αλλά ταυτόχρονα να δημιουργούνται και κάποιες, ε, κάποιες καταστάσεις οι οποίες ε, δημιουργούνται μερικές φορές μέσω των προβλημάτων στον ανταγωνισμό. Αν είσαι μια μεγάλη επιχείρηση ευρωπαϊκή, ακόμα και αν έχεις παγκόσμιες βλέψεις, ε, φυσικά θα πρέπει για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον ανταγωνισμό παγκόσμια πρέπει να είσαι σωστά εκπαιδευμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να ακούμε προσεκτικά τις επιχειρήσεις δηλαδή για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται ε, και ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι λεγόμενες νέες αγορές. Σχετικά με τις συγχωνεύσεις ε, αυτό το οποίο δεχόμαστε είναι ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συγχωνευτούν μπορούν να το κάνουν με την προϋπόθεση βέβαια ότι ε, εξακολουθεί να υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι ο μοναδικός δρόμος ε, που μπορούμε να ακολουθήσουμε αν πράγματι θέλουμε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός αν και υπάρχουν αρκετές διαφορές βέβαια ανάμεσα στις χώρες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός σε επίπεδο ευρωπαϊκό πάντα υπάρχει ένας πολιτής και πάντα υπάρχει ένας αγοραστής. Το θέμα είναι να δούμε πέραν αυτού τι μπορούμε να κάνουμε. Άνεμανς. Η νέα βελγική κυβέρνηση είναι πια στην τελική φάση σχηματισμού. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν προκύψει από την συνάδελφό σας την Μαριάν Τάισεν και φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα για την περίπτωση της τράπεζας Δέξια. Κάτι το οποίο αναφέρατε κιόλας και στις γραπτές σας απαντήσεις. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού βρήκε σε αυτή την περίπτωση ότι υπήρξε μια στρέβλωση ανταγωνισμού λόγω της ε, κρατικής επιδότησης. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Μιλάμε για 30 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το επίμαχο ποσό. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εσείς συγκεκριμένα, αποφασίσετε ότι πρόκειται για αποταμίευση και όχι για μετοχικό κεφάλαιο, αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για όλο το τραπεζικό σύστημα και την δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο Βέλγιο. Θέλω να θέσω το ερώτημα αυτό. Αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα. Ίσως είναι το τελευταίο θέμα που θα εμποδίσει τη δημιουργία μιας βελγικής κυβέρνησης. Ξέρετε κάτι γι' αυτό ή έχετε να σχολιάσετε ειδικά. Πρόεδρος ήθελα να σας διακόψει γιατί μακρηγορήσετε. Μπορώ όμως να σας δώσω λίγο χρόνο γιατί μπορώ να είμαι σύντομη στην απάντησή μου. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτα για αυτήν την υπόθεση. Λυπάμαι. Είναι ένα θέμα για, την, ε, για το σχηματισμό της βελικής κυβέρνησης και άμα δεν το ξέρετε και δεν ξέρει κανείς τίποτα γι' αυτό, χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Τότε όλα έχουν πάει καλά απόψε για σας, λέει η κυρία Βέσταγερ. Εντάξει, λέει ο Analyst Και πάλι. Σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, είναι λιγότερο από πέντε λιανοπολιτές που κυριαρχούν στην αγορά, λιανική αγορά τροφίμων στην Ευρώπη. 88, τη 88% της αγοράς καλύπτονται από τρεις τέτοιες εταιρείες στη Φιλανδία. Είναι φανερό ότι κυριαρχούν στην αγορά, εφαρμόζουν μεγάλο κόστος στην αλυσίδα παραγωγής και αυτό θίγει τους παραγωγούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αναπτυσσόμενες χώρες και υπάρχει και αντίκτυπος για τους καταναλωτές. Υπάρχει μια αποπτική αρχή για τα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει την ε, δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τρεις από τις τέσσερις όμως αυτές επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη. Χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση πώς θα μπορέσετε να εμποδίσετε τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσες θέσης. Πώς θα μπορέσετε να έχετε ισχυρούς εφαρμόσιμους κανόνες ώστε τα σούπερ μάρκετ να αντιμετωπίσουν με θεμητό τρόπο τους ε, προμηθευτές τους και τους καταναλωτές. Και πώς θα υπάρξει το ε, το θάρρος να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν πραγματικά να επιβιώσουν οι προμηθευτές και όχι να τους εξαναγκάζουν οι εταιρείες αυτές. Πράγματι ο ανταγωνισμός ιδιαίτερα στο λιανεμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται πάρα πολύ συχνά από τις εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό. Έχει σημασία να πούμε εδώ ότι όταν οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου λένε ότι αν το θέμα είναι γενικότερο τότε είναι και ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τον τομέα αυτό μόνο, ειδικά. Αλλά θα πρέπει οι ισχύουσες διατάξεις να εφαρμόζονται σωστά και στον τομέα αυτό και σε άλλους βέβαια. Θα ήθελα να, να θυμίσω εδώ η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής δημοσίευσε μια μεγάλη μελέτη για τον τομέα αυτό, μια μελέτη 400 σελίδων, την οποία βέβαια δεν πρόλαβα να διαβάσω ακόμα. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι προσπαθούν να κάνουν είναι να συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία για τις εμπορικές επιχειρήσεις, πόσες είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις, τι καινοτομία περιλαμβάνεται στα προϊόντα τα οποία πολλούν οι επιχειρήσεις αυτές, τι ρόλο παίζει η καινοτομία και χρησιμοποιούν την οικονομετρία για να αξιολογήσουν σωστά τον σωστό αριθμό των παικτών σε εισαγωγικά στον συγκεκριμένο τομέα. Βέβαια δεν είναι λύση μαγική, ε, έτσι και αλλιώς και η οικονομετρία έχει τα όρια της όπως ακριβώς και ο ανταγωνισμός. Αλλά νομίζω ότι ε, μπορούμε να βρούμε ε, κάποια στοιχεία θετικά, γιατί όπως είπα εδώ την πολλή δουλειά την κάνουν οι εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό. Θα το εξετάσουμε το θέμα ακόμα περισσότερο λόγω και της μελέτης όπως είπα η οποία κυκλοφόρησε σήμερα. Για την Ίνκο η κυρία Τούν und Höhenstein. Εδώ πίσω κάθομαι για να με δείτε. Θα συνεχίσω σε αυτή την ε, συζήτηση για τις κρατικές ενισχύσεις για την οποία εκφράστηκαν και τι ερωτήσεις. Μια συγκεκριμένη πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει τον καταναλωτή μέσω των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτού να επιλύσουν διασυνοριακές διαφορές. Αυτά τα κέντρα καταναλωτή ε, τα χρηματοδοτούν σε ένα βαθμό και τα κράτη-μέλη. Πρόσφατα ε, απεδείχθη ότι απερίφθη μια, προ... Ε, μια αίτηση για χρηματοδότηση ενός ε, κέντρου καταναλωτή γιατί η εθνική κυβέρνηση φοβήθηκε ότι μπορεί αυτή η χρηματοδότηση να κριθεί ως παράνομη κρατική ενίσχυση. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε αυτή η χρηματοδότηση που πάει στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτή δεν είναι όντως όχι κρατική ενίσχυση. Και επίσης, πολύ πιο γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα βιομηχανική πολιτική. Η βιομηχανία θα πρέπει να φτάσει στο 20% του ΑΕΠ το 2020. Ίσως λοιπόν θα πρέπει ορισμένα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να δούμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη τους χρειαστούν ή θελήσουν πιο χαλαρούς ε, κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Πώς εσείς μπορείτε Πώς μπορείτε λοιπόν εσείς να εξασφαλίσετε ότι θα επιβάλλονται σε σωστοί κανόνες παρά τις πιέσεις των κρατών μελών. Απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Να μην σταματάνε, να μην σταματάει η υποστήριξη από το φόβο ότι είναι παράνομη, ακόμα χειρότερα ασύμβατη με την ε, συνθήκη. Μα εάν προκύπτουν τέτοιε αμφιβολίε, μπορεί να διατυπωθεί το ερώτημα και να διευκρινιστεί με το τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη, όταν ε, πρόκειται για αυτά τα ζητήματα, να έχουν σαφείς και ισχυρές αρμοδιότητες. Ο εξυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων στον γενικό στον κανονισμό που προβλέπει τη γενική εξαίρεση, ε, δίνει τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη όχι μόνο σε ίσονο σημασία ζητήματα, αλλά σε πολλά θέματα να έχουν ε, μια παρέκκληση από τις κρατικές ενισχύσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και εμείς από πλευράς μας, από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε επαρκείς ε, πόρους για να διευκρινίσουμε εάν υπάρχουν ζητήματα, εάν πρέπει να υποβληθούν ερωτήματα και αυτή η κατανομή εργασίας θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί πότε πρέπει να βοηθήσουμε τον καταναλωτή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, πότε πρέπει να στηριχθούμε εμείς τον καταναλωτή ώστε να αμφισβητεί τις προτεραιότητες των κρατών μελών όταν πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις. Μια νέα διαφάνεια λοιπόν πιστεύω ότι χρειάζεται που θα προκύψει από τον εξυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Και είναι πολύ απαραίτητη γι' αυτό και στην προκείμενη περίπτωση έχουμε, πιστεύω, ανάγκη και από χρόνο και από πόρους όταν έρθει η ώρα να κρυθούν ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν τεράστιες ε, συνέπειες ως προς το τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια τα κράτη θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να διαχειρίζονται τους περιορισμένους πόρους του φορολογουμένου ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, έδειξε μια κάποια ανοχή για 10 δευτερόλεπτα κτλ. Ε, τώρα όμως θα σας παρακαλέσω να είστε πιο αυστηροί με το χρόνο γιατί πρέπει να τελειώσουμε στι 9. Η Σιάρο ο κύριος Λούκε. Ε, κυρία Βέσταγκερ, ε, απαντήσατε στην ερώτηση του κυρίου Μπάλτς ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να ε, μάλλον είπατε ότι θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να κρίνονται με τους ίδιους κανόνες ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο ε, ιδιοκτήτης τους, ποια, ποιας είναι. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, στο πλαίσιο της TTIP και η επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Όταν έχουμε δηλαδή από εδώ και μπρος να κάνουμε με αλλοδαπούς επενδυτές που επενδύουν στην Ευρώπη, οι εθνικές ρυθμίσεις μπορούν να καταστρατηγούνται και να μην υπάγονται αυτοί στα εθνικά δικαστήρια. Αυτό πιστεύετε ότι είναι στρέβλος του ανταγωνισμού και αν ναι πώς θα την αντιμετωπίσετε. Δεύτερον, όταν ένα ευρωπαϊκό κράτος επιβάλλει διόδια για την χρήση των οδών, του δικού του δικτύου, το οποίο, τα οποία διόδια αφορούν μόνο τους αλλοδαπούς χρήστες του οδικού δικτύου και όχι τους ημεδαπούς. Θεωρείτε ότι αυτό είναι παραβίαση του δικαίου περί ανταγωνισμού και αθέμητος ανταγωνισμός και άρα κατά των ευρωπαϊκών αρχών και ρυθμίσεων. Και αντιευρωπαϊκού πνεύματος επίσης. Δυστυχώς έχω περιορισμένη μονάχα γνώση για τα θέματα αυτά που λέτε σε σχέση με τις μεταφορείς. Αλλά πιστεύω ότι είναι ορθό να τεθεί το θέμα αυτό αν υπάρχει πράγματι διάκριση αν τα φορτηγά με ξένες πινακίδες πρέπει να πληρώνουν διόδια και τα φορτηγά με, εθνικά, με εθνικές πινακίδες όχι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ερευνηθεί, γιατί η απουσία διάκρισης είναι μία από τις βασικές αρχές, όχι μόνο της πολιτικής ανταγωνισμού, αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο είπε η Σεσίλια Μάλστρομ στη δική της ακρόαση για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, ήταν ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος και σαφής τρόπος να απαντήσει το ερώτημα αυτό. Υπάρχουν πολλές ιδέες, πολλές ανακοινώσεις που έχουν ε, διατυπωθεί. Υπάρχει η υποχρέωση να εξετάσουμε πραγματικά ποιος είναι ο κίνδυνος, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο φοβούνται πολύ ότι θα μπορούσε να συμβεί ποιες είναι οι ανησυχίες που υπάρχουν σε σχέση με την ε, επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσα τέτοια συστήματα ισχύουν ήδη σήμερα. Είμαι σίγουρη θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι ήταν κάπου 150.000 απαντήσεις οι οποίες ε, ε, βγήκαν από αυτήν την ε, διαβούλευση για τις ε, διαφορές μεταξύ επενδυτών και κρατών και ελπίζω ότι θα μπορέσω να διαβάσω κάποιες από αυτές τις απαντήσεις πρωτού επανέλθω στο θέμα αυτό. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να σας παραπέμψω στις απαντήσεις που έδωσε η Σίλια τη Δευτέρα για αυτό το θέμα. με την άποψή της. με την άποψη ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθηθεί από πάρα πολύ κοντά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διμερείς τέτοιες συμφωνίες οι οποίες δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Χρειάζεται λοιπόν μια ανοιχτή και πλήρης συζήτηση για την ισορροπία που πρέπει να εξασφαλιστεί. Ευχαριστώ η Σοφή Ιντβέλτ από την Άλτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βεστόε για την εισαγωγική σας ομιλία και την πάρα πολύ επιτυχή ε, απόδοσή σας στην διαδικασία της ακρόασης μέχρι τώρα. Ακούσαμε πολλά ήδη για τις πολιτικές ανταγωνισμού, ακούσαμε για την περίπτωση της ε, διαδικασίας antitrust κατά της Google. Τα προσωπικά στοιχεία είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της οικονομίας μας πια, αλλά η Κομισιόν μέχρι τώρα έχει βραδιπορήσει πάρα πολύ για να κατανοήσει ότι το big data, τα δεδομένα αυτού του είδου είναι πολύ πολύτιμα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Περιπτώσεις όπως τη Google, περιπτώσει που ακολούθησαν μετά την περίπτωση της Google, οι μονοπώλια μονοπόλια έχουν ε, αναπτυχθεί τα οποία δεν θα επιτρέπονταν ποτέ να υπάρχουν σε άλλους τομείς. Πολλές φορές η προστασία των δεδομένων παρουσιάζεται ως ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη του εμπόριου. Αυτό είναι σφάλμα. Στο παρελθόν η προστασία των δεδομένων ήταν στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά. Στι ΗΠΑ είναι αρμοδιότητα τη Federal Trade Commission. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά πράγματα η πολιτική ανταγωνισμού και η προστασία των δεδομένων. Αντί να αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό κατά περίπτωση και να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένε περιπτώσει στον πολιτικό στίβο, μήπω θα χρειαζόμασταν μια πιο πλήρη προσέγγιση για τους κανόνε ανταγωνισμού στην εποχή που έχουμε τόσο μεγάλη συλλογή δεδομένων. Θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μπορώ να αναγνωρίσω ότι το προφίλ των μεγάλων δεδομένων είναι το λεγόμενο νόμισμα του διαδικτύου. Έχουμε εδώ κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Όταν κάποιος έχει πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα ενός αλλά στα δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων, τότε μπορεί να κάνει αναλύσεις πολύ πιο διαφορετικές από αυτές τις οποίες ήταν ικανό να κάνει πριν από μερικά χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι προσπαθώντας να κατανοήσουμε ε, τον τρόπο που αναπτύσσονται οι αγορές αυτές. Δεν νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση και πώς μπορεί να συμβιώσουν από τη μία οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον ψηφιακό χώρο και από την άλλη με τα προσωπικά μας δεδομένα. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και νομίζω ότι και εσείς θα συνεργαστείτε, ελπίζω, με τις υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ε, το θέμα αυτό είναι ανάμεσα στον ανταγωνισμό και τα προσωπικά δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά το απότερο μέλλον, είναι κάτι το οποίο αφορά τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα δεν θα πρέπει απλά να συλλέγουμε στοιχεία αλλά να κατανοήσουμε ήδη από τώρα τον τρόπο που δουλεύουν οι αγορές και πρέπει η Γενική Διεύθυνση ε, για, τον, ε, για το εμπόριο να προσπαθήσει να κατανοήσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. κόφοντα. Ευχαριστώ. Είπατε ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ένα μοναχικό χαρτοφυλάκιο, αλλά είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με άλλα χαρτοφυλάκια. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Δανία και σε άλλες χώρες ίσως, είναι ότι οι επιδοτήσεις οι οποίες δίδονται σε ορισμένες επιχειρήσεις ναι μεν βοήθησαν τις επιχειρήσεις αλλά οι επιχειρήσεις αυτές κάποια στιγμή μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες ε, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι σημαντικό και ο Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό να είναι πολύ προσεκτικός έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις να μην χρησιμοποιούνται για την καταστροφή θέσεων απασχόλησης αλλά ε, με τα χρήματα αυτά να υπερασπιστούμε τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά λοιπόν χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και όχι για την καταστροφή. så, Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει πράγματι οι κανόνες να εφαρμόζονται με σωστό τρόπο. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις να παίρνουν επιδοτήσεις εάν έχουν σαν στόχο τα επόμενα χρόνια να μετακινήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μην βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους κανόνες. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να είμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολύ προσεκτικοί. Αν μια επιχείρηση λαμβάνει μια επιδότηση, ε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ποιους δίδουμε τα χρήματα, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα ευνοήσουμε συγχωνεύσεις και υπερσυγκεντρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Οι κανόνες λοιπόν θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί, αυτό είναι το βασικό. Εφόσον με επιβεβαιώσετε στη θέση του Επιτρόπου για τον ανταγωνισμό, και σε συνεργασία με τον αρμόδιο επίτροπο για τα περιφερειακά θέματα και για την εσωτερική αγορά, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για το θέμα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με ε, μοιρασμένη αρμοδιότητα και αυτό θα έλεγα θα χαρακτηρίσει και την αξιοπιστία και των επιδοτήσεων των ευρωπαϊκών, γιατί πράγματι πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι για την διευκόλυνση της μετακίνησής τους σε άλλες χώρες. Αυτό το ισχύει όχι μόνο για τον οικονομικό τομέα αλλά και για την έρευνα και για την καινοτομία κτλ. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ανταλάβουμε υπόψη μας προσπαθώντας να αξιολογήσουμε το σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Πρέπει να το βελτιώσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο Γεώργιος Κίρτσος από το ΕΛΚ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα τη γνώμη σας, όχι ως τεχνοκράτη, αλλά ως πολιτικού, για μία από τις μεγάλες προκλήσεις των, ε, για τις ευρωπαϊκές αγορές που προέρχονται από το τραπεζικό τομέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τεχνολογική τους υπεροχή, την εξαγωγική πολιτική της Κίνας, τα μεγάλα, τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, ενέργειας της Ρωσίας και την Gazprom, τα κρατικά μονοπόλια. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ε, απειλές, γιατί δεν μπορείτε βέβαια να ανοίξετε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα. Ο απερχόμενος επίτροπος ε, κύριος Αλμούνια, μεταξύ, στην τελευταία εμφάνιση του ενώπιον της Επιτροπής μας, μου φάνηκε ότι έχει παραδείχθει το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειές του και παρά την, ε, τις ικανότητες του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πολιτική της ισχύ, κάθε τύπου ε, ολιγοπόλια και μονοπόλια εξακολουθούν να ευημερούν. Ευχαριστώ. Αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά αν τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά δεν θα είχα και καθόλου δουλειά να κάνω εγώ. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιο. Κάποια από τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια. Οι αγορές δεν είναι τέλειες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανακαλύπτουμε συνεχώς ότι υπάρχουν μονοπόλια, ολιγοπόλια, τεράστιες επιχειρήσεις οι οποίες καταχρώνται των θέσεών τους στις αγορές και γι' αυτό θα πρέπει ε, η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού να είναι αυστηρή, δίκαιη, αλλά και στοχευμένη γιατί τις ορισμένες από τις αγορές τις οποίες αναφέρατε, η δύναμη του ε, καταναλωτή ε, δεν επιτρέπει πολλές αλλαγές. Και γι' αυτό ο καταναλωτής επαφίεται σε μας και εξαρτάται από μας, για να υπάρξουν σωστές αλλαγές. Ενέργεια, ψηφιακός κόσμος, χρηματοπιστωτικός τομέας εξαρτώνται από μας οι καταναλωτές έτσι ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να το πετύχουμε αυτό και ελπίζω να συνεργαστούμε και με την δική σας επιτροπή με τον καλύτερο τρόπο γιατί εσείς είσαστε κοντά στον κόσμο, στις, στους εκλογείς σας, στις περιφέρειές σας. Ακούτε πράγματα που δεν ακούω εγώ και γι' αυτό δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο μια επίσημη αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και μια αν θέλετε εμπειρική γνώση των προβλημάτων και να συζητάμε, όχι βέβαια τα απόρριτα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα θέματα τα οποία δημιουργούν ε, προβληματισμό. Έτσι θα περάσουμε σε μια πιο πλούσια και ελεύθερη Ευρώπη. Η κυρία Παούνοβα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κοιτάτε προς τα δεξιά, αλλά για κάποιο λόγο οι οργανωτέ τη συνεδρίας με βάλαν αριστερά παρά το γεγονό ότι ανήκω στο ΕΛΚ. Βέβαια κρατάω τη θέση κάποιων σοσιαλιστών που λείπουν απόψε. Βλέπω ότι έχουμε το ίδιο πάθο για σοκολάτα. Ελπίζω ότι θα βρούμε και κοινό έδαφο σε άλλου χώρου. Όπω ξέρουν πολλοί από εσά, η υπεράπτωση τη ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι μια από τι βασικέ μου προτεραιότητε σε επίπεδο πολιτική. Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν να δώσουμε τα σωστά κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων υψηλή προσθέμενης αξία, ιδίω για τη νέα γενιά στον τομέα τη ψηφιακή ενωμένη αγορά. Πιστεύω ότι η βιομηχανία πληροφορική και επικοινωνία είναι από του κύριου μοχλου για να επιτύχουμε αυτού του στόχου. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η προσέγγισή σας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του ψηφιακού θεματολογίου στην πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε ότι η παρέμβαση του δικαίου του ανταγωνισμού μπορεί να είναι ε, αρνητική στον τομέα αυτό λόγω της ταχείας εξέλιξης στον τομέα αυτό και μήπως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν παρεμβαίνουμε σε θέματα σχεδιασμού προϊόντων. Λυπάμαι, λέει ο πρόεδρος. Και διακόπτει την ομιλήτρια. Και αυτή η σοκολάτα προέρχεται από μια πολύ καλή συγχώνευση. Είναι ε, γλυκάνισος μαζί με με, με, με μαύρη σοκολάτα. Μα δεν έχουμε μόνο το κοινό πάθος σοκολάτα. Έχουμε και το πάθος να δημιουργήσουμε θέσεις υψηλής προσθέμενης αξίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσει η Ευρώπη να βρει μια σωστή θέση στην αλυσίδα παραγωγής προσθέμενης αξίας και να μπορέσει να αλληλεπιδράσει με θετικό τρόπο με την παγκόσμια οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι μονάχα να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία, αυτή καθεαυτή, αλλά να, να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε και εμείς μια σωστή θέση σε αυτή την αλυσίδα και παράγουμε αξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο χώρος της πληροφορικής είναι πάρα πολύ σημαντικός από αυτή την έποψη. Εγώ πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός αυξάνει την καινοτομία και η εφαρμογή κανόνων antitrust θα ενισχύσει και, και αυτή η εφαρμογή την καινοτομία. Γιατί αν έχετε πολύ μεγάλες εταιρείε οι οποίες κυριαρχούν απόλυτα στον τομέα της πληροφορικής, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να φέρουν τις καινοτομίες τους στην αγορά. Αν δεν εφαρμόζονται οι κανόνες αντιτράστ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δει καταπληκτικά παραδείγματα πάρα πολύ μικρών εταιριών οι οποίες δεν θεωρούν καν ότι είναι εθνικές εταιρείες. Από τα γενοφάσκια τους θεωρούν ότι είναι παγκόσμιες εταιρείες ακόμα και αν έχουν δύο ή τρία άτομα που δουλεύουν και σε ένα πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα γίνονται παγκόσμιες. Δεν έχουν περάσει από μια φάση προάσπισης και προστασίας από τα κρατημέλη. Κανείς δεν τις ε, να νούρισε για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Απλώ επειδή έχουν πολύ καλέ ιδέε μπορέσαν να φτάσουν σε επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την Επιτροπή η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές είναι οι θέσεις και από την πλευρά του ΕΛΚ, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση. Κύριε υποψήφια, Επίτροπε, τι μέτρα συγκεκριμένα σκοπεύετε να θεσπίσετε ώστε μηχανισμό συλλογική επανόρθωση σε περίπτωση παραβιάσεως των κανόνων ανταγωνισμού ε, να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί. Πιστεύετε ένα τέτοιο συγκεκριμένο μηχανισμό θα πρέπει να ενσωματωθεί σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό συλλογική συλλογικής επανόρθωση οριζόντιο και πιο συμπεριληπτικό και τι μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε προκειμένου να προστατέψετε τα δικαιώματα των καταναλωτών, ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζοντάς τους και ευρύτερε επιλογές και αν πρόκειται να αντισταθείτε στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσετε μια ισότιμη μεταχείριση, μη διακριτική, ισοδίκαια έναντι των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην ιστορική αγορά. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, με μεγάλη ε, χαρά διαπίστωσα, ήταν ευχάριστη έκπληξη, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον ανταγωνισμό η συνήθις διαδικασία, η νομοθετική διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζεται όταν μιλούμε για ζητήματα επανόρθωσης ή αποζημίωσης. Από τον ε, κύριο Αλμούνια και συλλογικά από την Επιτροπή έχω ενημερωθεί ότι υπήρχε η αντιμετώπιση κατά τρόπον συνεργατικό με το Συμβούλιο, ιδιαίτερο και με το Κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερο για το αποτέλεσμα που προέκυψε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τη δική του ιστορία ήδη, αλλά θα χρειαστεί να το ξαναδούμε σε κανένα δύο χρόνια όταν έχουμε μια εικόνα για το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω, διότι όταν έχουμε να κάνουμε με αποκατάσταση ζημίας. Μπορούμε να έχουμε μια διτή προσέγγιση έναντι των εταιριών που δεν τηρούν τους κανόνες και την επιβολή του νόμου από την Επιτροπή και την ιδιωτική επιβολή. Δηλαδή, εάν ε, κάποιος παραβιάζει τους κανόνες, τότε πρέπει να πληρώνει και το δυσχετικό τίμημα. Τα πρόστιμα ε, που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από την Επιτροπή έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά τους, δηλαδή πόσο ζημιώσαν την αγορά. Όταν όμως έχουν ζημιώσει καταναλωτές, τότε επιβάλλονται ακόμη επιπλέον πρόστιμα, συμπληρωματικά δηλαδή, και πρέπει να είναι πιο βαριά ακόμη. Αυτό είναι ο αποτρεπτικός ρόλος που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε για τα πρόστιμα αυτά, διότι μόνο με καλή, ανοιχτή αγορά και ισότιμη ε, στάση των επιχειρήσεων μπορούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Άρα θα είμαστε και πολύ διεξοδικοί στην έρευνα, στη διερεύνηση και θα ε, φροντίσουμε τα, προφι, τα πρόστιμα να είναι υψηλά ώστε να μην μπορούν απλώς να εκφράσουν μια γραμμή του ισολογισμού ε, σαν έξοδα της επιχείρησης, αλλά να αντιστοιχούν στα κέρδη που έχουν εξασφαλίσει από την αθέμητη συμπεριφορά και να είναι πραγματικά αποτρεπτικά. Η κυρία Ρίνα Κάρη, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω για το πρώτο τουλάχιστον κομμάτι της ερωτήσεώς μου στο θέμα του ανταγωνισμού και του κοινωνικού dumping που ακούστηκε νωρίτερα. Ξέρετε και εσείς ότι στη Δανία έχουμε ένα σύστημα βάσει του οποίου καταχωρίζονται σε, έναν, σε ένα μητρό οι ελοδαπές επιχειρήσεις και έτσι οι ε, υπηρεσίες, οικονομικές, φορολογικές επιχειρήσεις και τα συνδικάτα ακόμα μπορούν να επαληθεύουν τι στάση έχουν αυτές οι επιχειρήσεις σε σχέση με την τήρηση νομοθεσίας, εάν δίνουν μισθούς σωστούς, εάν τηρούν τις κοινωνικές προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να το επαληθεύσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως, διάβρο, ως τρέβλωση του ανταγωνισμού. Έχει ήδη πει η Επιτροπή ΔΕ ότι θα παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή με το μητρό αυτό της ε, Δανίας. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο μπορείτε να υπερασπιστείτε σαν λύση ή μπορεί να κινδυνεύουμε να το δείτε ως στρέβλος ανταγωνισμού απάντηση. Εγώ πάντοτε θα μεριμνώ να είναι οι συνθήκε συμμετοχής στην ε, δραστηριότητα της αγοράς ισότιμας. Δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό ο οποίος συνεπάγεται όλο και χαμηλότερες προδιαγραφές. Πρέπει να είναι υγιή ο ανταγωνισμός. Αυτό το μητρό που υπάρχει στην Δανία βεβαίως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά βεβαίω και μπορεί να συζητηθεί το αν είναι ενδεχομένως υπερβολικό σε αυτό που κάνει. Ένα μητρό δηλαδή το οποίο δεν λέει μόνο ποιος είναι εγκατεστημένος, έχει την έδρα του στην χώρα και τι δραστηριότητες αναπτύσσει, ε, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα μητρό το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να είναι πολύ βαρύ γραφειοκρατικά και μπορεί να αποθαρρύνει κάποια επιχείρηση να μην ε, τολμήσει δηλαδή να έρθει να εγκατασταθεί στην ε, Δανία, να αναπτύξει δραστηριότητε, γιατί αυτό θα σήμαινε πολύ σημαντική γραφειοκρατική επιβάρυνση λόγω του Μητρώου κτλ. Εάν πρόκειται για αλλοδαπή επιχείρηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να βρούμε λύσει. Οι κανόνε του ανταγωνισμού φυσικά πάντοτε θα τιμωρούν εκείνου που καταστρατηγούν τι συνθήκε του ανταγωνισμού. Αλλά αν κάποιο έχει μια ευκαιρία με ένα καλό προϊόν να προσφέρει στην αγορά, να πουλήσει το προϊόν του στην αγορά να προσφέρει μια υπηρεσία, δεν πρέπει να τον εμποδίσουμε. Ευχαριστώ, Μάικ Ραϊμόν Πράσινη κυρία Επίτροπε, για τον ανταγωνισμό σε φορολογικό επίπεδο. Έχετε δώσει μια διπλωματική ίσως ε, απάντηση. Εντάξει, καταλαβαίνω πρέπει να είστε διπλωματικοί και να δείχνετε προσοχή στα θέματα αυτά. Η Γενική Αντιπρο... Διεύθυνση Ανταγωνισμού έδωσε στοιχεία για ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες στην Ιρλανδία, στις κάτω χώρες και στο Λουξεμβούργο. υπήρξαν κάποιες ε, διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά με τις εταιρείες αυτές. Η πρώτη κρίση της Κομισιόν είναι ότι αυτές οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί με τις χώρες αυτές και τις πολυεθνικές εταιρείες είναι, πολύ, είναι παράνομες κρατικές επιδοτήσεις. Ξέρω ότι δεν υπάρχει ακόμα μια οριστική απάντηση μέχρι ότου έχει γίνει πλήρης διερεύνηση αυτής της υπόθεση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η πολιτική σας κρίση για το θέμα αυτό και εάν έχετε κάποια περαιτέρω σχόλια για τις υποθέσεις αυτές. Αυτό το οποίο θέλω είναι αν υπάρχει κάποια υπόθεση πρέπει να την κερδίσουμε στα δικαστήρια να την κερδίσουμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα έχουμε τις αποδείξεις και θα μπορούμε να τεκμηριώσουμε αυτές τις υποθέσεις, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα που θα δώσουμε στις άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αν υπάρχει πράγματι μια τεκμηριωμένη υπόθεση εναντίον αυτής της φοροαποφυγής, εναντίον αυτών των εταιριών που μπορούν να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες για να μην πληρώνουν το φόρο που θα έπρεπε να πληρώνουν. Και από τη έχω δει μέχρι στιγμή, τα πράγματα αυτά είναι πολύ πλοκά. Δεν είναι θέμα μοναχα κανόνων, είναι θέμα και <clears throat> κρίσεων των δικαστηρίων. Γι' αυτό θα πρέπει να μπούμε σε πολύ μεγάλο βάθος σε αυτή την έρευνα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα σταθερό έδαφος επί του οποίου να βασίσουμε αυτή την υπόθεση. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να ευδοκιμήσει στο δικαστήριο μια τέτοια υπόθεση εναντίον των εταιριών αυτών και των κρατών. Νομίζω ότι η προτεραιότητά μας και η φιλοδοξία μας είναι να το πετύχουμε αυτό. Αυτό δεν έχει σαν στόχο να οδηγήσει από την πίσω πόρτα την Ευρώπη σε μια κοινή φορολογική πολιτική. Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να έχει διαφορετικά επίπεδα φορολογίας επιχειρήσεων στο ε, άμεσο μέλλον. Υπάρχει αυτή η πρόταση για μια εδρεωμένη φορολογική βάση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η λύση για όλα αυτά τα προβλήματα. Βασικά όμως πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να έχουμε τους πόρους για να το πετύχουμε και αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό, ενδεχομένως μπορούμε να το κάνουμε σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο να είναι πεπερασμένο και να μην κρατάει μέχρι το τέλος του κόσμου. Βερόνικα Λόπεθ Φοντανιέτ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, έχει πολύ μεγάλη σημασία το χαρτοφυλάκιό σας και οι ρυθμίσεις που αφορούν το χαρτοφυλάκιο απαιτούν, θα έλεγα, απαιτείται μάλλον να εφαρμόζονται με σωστό τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ε, με δίκαιο τρόπο κατανομή όλων των ευθυνών. Να αναφερθώ τώρα στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, σημαντικό τομέα για την τεχνολογία, την οικονομία και την απασχόληση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει τον τομέα αυτό με τον πιο δίκαιο τρόπο. Ξέρετε για τις καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει εις βάρος των, της εταιρείας Γέρος Εσπανιόλες σχετικά με κάποιες α, ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στη μία περίπτωση και δεν έγιναν στην περίπτωση των Ολλανδικών ναυπηγείων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν εσείς θα δεσμευτείτε να εφαρμοστεί ε, δίκαιος τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των θεμάτων που άπτονται της κοινοτική νομοθεσίας. Δεν ξέρω ε, καθόλου θα έλεγα την υπόθεση αυτή σχετικά με την ε, βιομηχανία την αυπηγική. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά γενικότερα και υπάρχει παγκόσμιος ανταγωνισμός. Οι μεταφορές ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές έτσι και αλλιώς για το σύνολο της οικονομίας και πέραν αυτού έχει σημασία και ο συγκεκριμένος τομέας να σέβεται τους κανόνες του ανταγωνισμού και έχει μεγάλη σημασία όταν υπάρχουν υπο, υποψίες ότι κάποιες άλλες ε, ε, νομικές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο ε, σε άλλη χώρα είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα. Και το κόστος της μεταφοράς γενικότερα εξαρτάται από το αν μπορεί κανείς να αναφυγήσει σκάφη και με την βοήθεια κρατικών επιδοτήσεων. Ο κύριο Τζάνι, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσετε. Η προκάτοχό σας είχε ξεκινήσει πάρα πολλές έρευνες, χωρίς όμως το τέλος να καταλήγει σε συμπεράσματα. Ε, πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε εσείς, θα υπάρξει αλλαγή ή θα συνεχίσουμε αυτά τα οποία έκανε ο Αλμούνια. Δεύτερον, για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων. Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών πολλές φορές αγνοούνται και θίγονται οι μικρομέτοχοι και υπονομεύεται η αξία των επενδύσεών τους υπέρ μάλιστα αυτών οι οποίοι λειτουργούν με διαφορετικό καταχρηστικό τρόπο. Πώς θα προστατεύσετε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων μικρομετόχων Για το τελευταίο θέμα, ε, είναι κάτι το οποίο άμεσα οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν εξασφαλίζουν βέβαια. Όταν ε, ε, μελετάτε μια συγχώνευση πολλά θέματα θα πρέπει να εξεταστούν για τον πώς θα λειτουργήσει η νέα εταιρεία, αν θα υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά στην οποία ε, θα ε, μπει η εταιρεία αυτή. Και ε, κάποια από τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνονται και αυτά τα οποία είπατε εσείς. Μπορώ να ακούσω το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας όμως, λέει η κυρία Βέσταγκερ, γιατί απαντώντας το δεύτερο ξέχασα το πρώτο. Ευχαριστώ κύριε Σάφη. Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον επόμενο ε, Ήταν για την προσέγγιση της δουλειάς σας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, τις έρευνες, ακόμα και αν δεν καταλήξουν σε πρόστιμο. Αλλά να μπορούμε να ερευνήσουμε αν πρόκειται για καρτέλ, ε, η συγχώνευση ή παραβίαση του νόμου κατά τον, ε, του αντιτράστη, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν είναι υποχρεωτικό όμω να επιβληθούν οι σχετικέ κυρώσει, γιατί αν είναι έτσι δεν αρχίζουμε καν. Και άρα περιορίζουμε πολύ το πεδίο δράση μα. Είναι σημαντικό λοιπόν, πιστεύω, να έχουμε διακρατική ευχέρεια και να βεβαιωνόμαστε ότι όταν υπάρχει και υποψία θα διερευνηθεί για να αποδειχθεί έστω και μετά ότι δεν ήταν βάσιμη. Αυτό πρέπει να μπορούμε να το δεχθούμε. Και ως εκ τούτου θα πρέπει ίσως κάποιες διαδικασίες του, που έχει ανοίξει ο Επίτροπος Αλμούνια να συνεχιστούν. Πάντως σημαντικό είναι να έχουμε αρκετά ταχείες διαδικασίες. Γιατί είναι σημαντικό για μια επιχείρηση ή να είναι τομέα ακόμα, αν βρίσκεται υπό έρευνα, να λάβει γρήγορα μια απάντηση, ειδικά όταν αυτή είναι αρνητική. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Σάντλ Μοζέ, εκ μέρους Επιτροπής της Ιστορικής Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ, Μαγκρέτε. Θέλω να σου πω ότι ασφαλώς και δεν είναι πολύ γραφειοκρατικό αυτό το μητρό για το οποίο έγινε κουβέντα νωρίτερα για την ε, ε, δανεία. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να εφαρμόζονται. Βεβαίως χρειάζονται και άλλα μέσα ίσως, ε, ώστε να έχουμε πιο καλή, την ιδανική θα έλεγα, ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν Ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπιστεί μια επιτροπή, μια ομάδα ε, task force η οποία θα ταξιδεύει ανά την Ευρώπη και θα ψάχνει να διερευνήσει υποθέσεις ε, παραβίασης του ανταγωνισμού. Ε, παραδείγματι άμα διαπιστώνεται παραβίαση των τιμών των κανόνων περί τιμών, αν εμφανίζονται συνθήκες καρτέλ κτλ. Εσείς θα υποστηρίζετε μια τέτοια πρόταση στην Ευρώπη. Απάντηση. να, αυτό είναι, ας πούμε, μία από τις προτάσεις που κανείς θα μπορούσε να ξανασκεφτεί προσεκτικά. Αυτό βέβαια είναι τι είδου ε, αντίκτυπο θα έχει το έργο μια, απο τις προτασεις που κανεις θα μπορουσε να ξανασκεφτει προσεκτικα αυτο βεβαια ειναι τι ειδου ε αντικτυπο θα εχει το εργο μια τέτοια μιας τέτοιας ομάδας ή task force. Αλλά βεβαίως και θα πρέπει να κοιτάμε πράγματα συγκεκριμένα και οι γενικέ ευθύνσει τη υπηρεσία. θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν συγκεκριμένες καταστάσεις και να λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Και γι' αυτό είναι σημαντικό επίσης να εμφανίζονται τα μέλη του προσωπικού για να διερευνούν υποθέσεις επιτόπου όπου υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλά αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό της δουλειάς των εθνικών ε, εποπτικών αρχών του ανταγωνισμού και σε συνεργασία μαζί τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, αυτές οι υπηρεσίες οι εθνικές έχουν πνεύμα ε, ανοιχτό και προς τα ευρωπαϊκά θέματα ή μπορεί να δοθεί καλύτερα η λύση των προβλημάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αλλού μπορεί οι εθνικές αρχές να έχουν πολύ καλύτερη θεώρηση για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στη χώρα. Η υπηρεσία, η δανέζικη, η βουλγάρικη, η ισπανική μάλλον γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση στα θέματα του ανταγωνισμού μέσα στη χώρα της. Και γι' αυτό θα πρέπει ε, να φροντίσουμε να μπορούμε να εμπιστευθούμε και τις εθνικές αρχές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συσταθεί μια μεγάλη ομάδα που θα ταξιδεύει δεξιά στην Ευρώπη. Οι εθνικές αρχές μπορούν να μας ενημερώνουν πολύ καλά και έγκριτα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ Μάρκους Μπρέτσελ, Ίμκο και πάλι, ECR, στετικοί μεταρρυθμιστές. Κυρία Βέστεγερ. Το 2013 έγινε η πρώτη ε, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών κατά της ε, ιδιωτικοποίησης του ύδατος, των, ε, της υδροδότησης και επομένως της εξαίρεσης από την οδηγία του ύδατος. Υπήρξαν πολλές λοιπόν κινήσεις ε, προς την κατεύθυνση αυτή και το θέμα αυτό του της ιδιωτικοποίησης των υδάτων πόρων είναι κάτι το οποίο εμπεριέχεται στη διαπραγμάτευση συμφωνίας TTIP με την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξαν μικτές εμπειρίες από τη δημιουργία μονοπωλίων στον τομέα αυτό και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για τη δυνατότητα φυσικά μονοπόλια να ιδιωτικοποιηθούν και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίζατε, θα αντιμετωπίζατε τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ιδιωτικό μονοπόλιο στα, στα θέματα του, της υδροδότησης και ποια είναι η στάση σας σε σχέση με τις προσπάθειες στο, στη συμφωνία TTIP να επιβληθεί ένα τέτοιο μονοπόλιο σε ιδιωτικό επίπεδο για το νερό. Πρώτα απ' όλα, λέει η κυρία Βέστοερ, οι πρωτοβουλίες των πολιτών. Νομίζω ότι ήταν ορθές. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μια πρωτοβουλία πολιτών. Όχι μόνο αυτές οι οποίες φτάνουν το κατόφλι το ενός εκατομμυρίου υπογραφών, αλλά και αυτές που ξεκινούν στη βάση και αλλάζουν την οτροπία γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε αυτό το νέο εργαλείο στη δημοκρατία μας, την, της πρωτοβουλίας των πολιτών και πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει και την ευρωπαϊκή συζήτηση για τα θέματα αυτά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στο θεσμικό τρίγωνο Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου. Τώρα όταν πρόκειται για φυσικά μονοπόλια και την ιδιωτικοποίησή της δεν ξέρω αρκετά πράγματα για τις διαπραγματεύσεις στο επίπεδο της συμφωνίας TTIP και αν πράγματι θα επηρεάσει τα πράγματα για να αντιμετωπίζω το ερώτημά σας σε συγκεκριμένο επίπεδο. Μπορώ να επανέλθω όταν μάθω περισσότερα βέβαια. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Ο Μάκελ Φόρια για την Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Βεστάκερ, στις σας ερωτήσεις, στις ερωτήσεις μας. Αναφερθήκατε στην κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στην πρακτική, πολύ συχνά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, υποφέρουν από την γραφειοκρατική επιβάρυνση της έγκρισης ή των συνθήκων ε, για το περιβάλλον. Πολλές είναι επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες, οι οποίες ε, ταλαιπωρούνται και υποφέρουν από τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν στα διάφορα κράτη ευρωπαϊκά εκατομμύρια. Εάν λοιπόν θέλω ε, ένα ε, δάνειο του ύψους των 50 εκατομμύριων, το οποίο δεν είναι βέβαια και μικρό, είναι για τις mid-cap όμως σημαντικό, τότε έχουμε 25 εκατομμύρια επιβάρυνση. Θα ήθελα να ρωτήσω τι είδους δυνατότητα δράσης μπορεί να έχει μία ε, επιχείρηση και πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε από τη θέση σας ως Επίτροπος Ανταγωνισμού. Απάντηση. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Τρία χρόνια ήμουν αρμόδια για θέματα οικονομίας και εσωτερικών ως υπουργός της πατρίδας μου και είδα ότι χρειάζεται και οι επαγγελματίες να έχουν περισσότερο περιθώριο και λιγότερο, λιγότερη γραφειοκρατία. Γιατί πρέπει όχι μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οι δημόσιοι φορείς να βρουν ε, περιθώριο δράσης. Είναι ένα θέμα λοιπόν πολύ σημαντικό που έχουμε έναν πρώτο αντιπρόεδρο επικεφαλής και Βεβαίω δεν θα άφηνα το θέμα στην αρμοδιότητά του, θα ήταν και σωστό, αλλά θα συνεργαζόμουν μαζί του για την αποδιάρθρωση της γραφειοκρατίας ή για λύσεις που θα σήμαιναν ότι η μελλοντική νομοθεσία θα έδινε απλούστερες ε, απαντήσεις στα προβλήματα. Μια ισορροπία ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπώνεται η νέα, η νέα νομοθεσία, ώστε να είναι σκόπιμη και η αρμόζουσα ε, λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο ε, αντί να επιλύεται με 28 διαφορετικές νομοθεσίες, επιλύεται από μία ευρωπαϊκή. Και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε στο πώς διατυπώνεται αυτή η νομοθεσία, πώς ε, ε, εκπονείται αυτή η νομοθεσία, για να μην προσπαθεί κανείς να το παρακάνει όπως θα λέγαμε, δηλαδή να έλεγε «Α, να, μια στιγμή έχουμε το νομοθέτημα, αλλά ας βάλουμε και λίγες στατιστικές μέσα, ας βάλουμε και κανένα δύο διατάξεις παραπάνω και τελικά να φτάνουμε στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα». Εμείς θα λέγαμε το ανάποδο λοιπόν. Αντί να ζητάμε όλο και πιο πολλές διατάξεις, όλο και πιο πολλές ρυθμίσεις, να κοιτάγαμε ποιες είναι οι ελάχιστες απαραίτητες. Και ως ρυθμιστές βεβαίως μπορούμε να αξιοποιούμε υφιστάμενα ε, δεδομένα και να μην ζητάμε από την επιχείρηση να μας διαθέτει όλο και ε, να μας διαθέτει κάθε φορά τα ίδια δεδομένα για τις ε, στατιστικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε νομίζω να ε, κοιτάξουμε μεγάλη προσοχή γιατί θα είναι κρίσιμε σημασία για τον τρόπο με τον οποίο εκπονείται η νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο Μάρκους Φέρμπερ αντιπρόεδρος και νέος πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Επιτροπής μας για τον ανταγωνισμό. Ένας τρόπος που βρέθηκε από πλευράς μας για να αναβαθμίσουμε τις πολιτικές ανταγωνισμού με την ελπίδα ενός επικοδομητικού διαλόγου με την νέα Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό, ε, ο κύριος Φέρμπερ. Βεβαίως, αν, προσφέρετε, αν μου λέτε ιδέες για καφεδάκι, πολύ ευχαριστώ να τις αξιοποιήσω, αλλά μπορούμε και κανένα ποδοσφαιρικό αγώνα μαζί. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια είχαμε μεγάλες υποθέσεις ε, αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ε, ανταγωνισμού με μεγάλε επιχειρήσει και κυρίω διαδικτύου όπω η Google. Πιστεύετε λοιπόν ότι οι ρυθμίσει που υφίστανται αυτή τη στιγμή στο δίκαιο του ανταγωνισμού είναι οι αρμόζουσε για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν στην ψηφιακή οικονομία. Εάν όχι, ποιε θα πρέπει να είναι οι καινούριε ρυθμίσει. Και δεύτερον, υπάρχει ένα ζήτημα δικαίου του ανταγωνισμού, μια σύμβαση δηλαδή, μια συνθήκη μάλλον ε, ε, συνεργασία στο δίκαιο του ανταγωνισμού με την Ελβετία. Ε, όπου προβλέπεται να υπάρξει ανταλλαγή στοιχείων χωρίς να ενημερώνει το ενδιαφερόμενος. Πώς βλέπετε αυτή τη συμφωνία με την Ελβετία και θεωρείτε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σύναψη περαιτέρω συνθήκων και αν ναι με ποιες χώρες. Όλα αυτά είναι πολύ καλά ερωτήματα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε περαιτέρω. Αν σα φέρω καφέ θα μου φέρετε λοιπόν πιο πολλά ουσιαστικά στοιχεία για τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ οι αλλαγές που μπορούμε να δούμε πόσο έχουν αλλάξει οι αγορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να σας ε, υπενθυμίσω πώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν όταν ήταν οι δίσκοι μακράς ή οι μηχανές φαξ κτλ. Είναι δύσκολο λοιπόν να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αυτή είναι η πρόκληση ενώπιόν μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να ε, καταχραστεί μιας δεσπόζουσας θέσης, ότι μια, ε, ότι μια συγχώνευση πρέπει να αφήνει άθικτο ακόμα τον ανταγωνισμό όσο πιο πολύ μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω ότι αυτά τα παλαιομοδίτικα πράγματα εξακολουθούν πολλά από αυτά να έχουν μια εγκυρότητα. Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και να δούμε τι γίνεται στις καινούργιες αγορές, στις ψηφιακές. Αυτό είναι πραγματικά μια πρόκληση. Σε ορισμένε περιπτώσεις που τώρα είναι υπό εξέταση εμφανίζονται συνέχεια νέα στοιχεία. Όχι καθημερινά, αλλά κάθε μια-δύο εβδομάδες βγαίνουν και νέα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα τέχνασμα για να α, καθυστερήσει η απόφαση, γιατί κάποιες αποφάσεις πρέπει εν καιρό να ληφθούν. Η συμφωνία με την Ελβετία έχει κάπως ειδικό χαρακτήρα. Είναι από τις λίες τέτοιε τέτοιες συμφωνίες που έχουν και το στοιχείο αυτό της ανταλλαγής πληροφοριών. Και θα ήθελα να συζητήσω και μαζί σας πώς θα πρέπει να διαμορφώνται συμφωνίες αυτού του είδους, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι συμφωνίες, γιατί θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Από αυτά τα οποία έχω μάθει, υπάρχει πολύ καλή σχέση εργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανικών αρχών. Αυτό είναι πολύ θετικό. Και επίσης με τις Καναδικές αρχές έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Πιστεύω ότι ένα διεθνέ δίκτυο αρχών ανταγωνισμού θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο εποπτεία του ανταγωνισμού. Και μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε και σε θεματικό επίπεδο τη λειτουργία αυτών των δικτύων. Ο Σβέν Γκίγκολτ για τους πράσινους έχει το λόγο τώρα. Κυρία Βέστρια, τα τελευταία χρόνια. Ο τομέας όπου έχουν αυξηθεί περισσότερο οι κρατικές επιδοτήσεις είναι οι τράπεζες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν διασωθεί τράπεζες με δημόσια χρήματα. Η τελευταία Κομισιόν το είχε εγκρίνει αυτό, αλλά αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο με τον τρόπο αυτό έχει την προοπτική να αλλάξει. Υπήρξαν πολλές πιέσεις που ασκήθηκαν από ορισμένα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ε, περίπτωση αυτή των ε, βοηθειών και τη μείωσή τους, ιδίως στη φάση αυτή των ε, τεστ δοκιμασίας αντοχής. Εσείς υποστηρίζετε τέτοιου είδους αρρώγειας. Δεύτερον υπάρχει το, η διαμαρτυρία ότι δεν υπήρξαν σαφή κριτήρια για το ποιος διασώθηκε και πώς και για την ε, συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία αυτή, ότι έγινε με αδιαφανή τρόπο. Εσείς λοιπόν είσαστε ε, έτοιμοι να διευκρινίσετε και να ερευνήσετε τι ακριβώς έχει γίνει για όλες αυτές τις τράπεζες οι οποίες ήταν αποδέκτες ποσών για να διασωθούν. Well, you are σωστό αυτό. Προφανώς Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε ότι υπήρξε μία προσπάθεια ανταπόκρισης στην κρίση. Και έγιναν προσπάθειες να ξεφύγουμε από το πρόβλημα και να περάσουμε σε ένα χρηματοπιστωτικό τομέα πιο υγιή. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχουν θέματα κρατικών επιδοτήσεων εδώ, ακόμα και όταν τεθεί σε λειτουργία συνολικά το, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Και θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν προβλήματα όταν δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου της αντοχής τους και υπάρχουν τράπεζες οι οποίες θα έχουν ανάγκη περισσότερα κεφάλαια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι τίθεται το θέμα της κρατικής επιδότησης. Υπάρχουν νέοι κανόνες, υπάρχει βέβαια εξυγχρονισμός αυτού του τύπου της βοήθειας προς τα πιστοτικά προβλήματα. Ε, περάσαμε, φτιάχνουμε μια γέφυρα από το bailout προς το bail-in όταν τεθεί σε λειτουργία η Τραπεζική Ένωση. Τώρα είμαστε σε μια ενδιάμεση αν θέλετε περιοχή και γι' αυτό θα πρέπει οι κανονισμοί για την κρατική βοήθεια να λειτουργούν σωστά ε, μετά από τα αποτελέσματα ε, των stress test στο τέλος του μήνα. Η έρευνα. Δεύτερη ερώτηση δηλαδή. Ναι, Δεν έχω μια γενικότερη άποψη ακόμα για αυτούς οι οποίοι ωφελούνται. Δεν γνωρίζω ακόμα πώς μια τέτοια έρευνα ε, θα εξελιχθεί και τι θα καλύψει. Ξέρω ότι τα διάφορα κράτη έχουν λειτουργήσει διαφορετικά. Κάποια έχουν προχωρήσει με τη μέθοδο της ανάκτησης των πιστώσεων αν τα πράγματα πάνε καλά. Άλλες ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές θα πρέπει να δω τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη μεμονωμένα έτσι ώστε να ελέγξουμε αν πράγματι υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε μια ιστερότερη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Βάλει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία μεση ερώτηση και μετά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχάς πώς μπορούμε να δώσουμε εγγυήσει στον ανταγωνισμό σε ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ πολυπίκυλο θα έλεγα και ευνοεί τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Η Fiat Chrysler μετέφερε το αρχηγείο της στην έδρα της ε, ε, τη διοικητική στην Ολλανδία, τα φορολογικά της στην Μεγάλη Βρετανία γιατί έτσι τη βολεύει ε, και στην Ιταλία κρατά ελάχιστα πράγματα. Ένας μικρός επιχειρηματίας δεν μπορεί να το κάνει αυτό για να ωφεληθεί από αυτές τις ρυθμίσεις. Οι μεγάλες οι μπορούν να το κάνουν αυτό και ωφελούνται από την απελευθέρωση των αγορών και από την πλήρη αυτή απορρίθμιση. Θέλω την αξιολόγηση τη δική σας για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν γνωρίζω την συγκεκριμένη περίπτωση. Uh, Αλλά αν ήμουν μια μικρή επιχείρηση, αυτό που έχει σημασία είναι οι ελεγκτικές και εφαρμοστικές αρχές να χρησιμοποιούν τις αρμοδιότητές τους. Γιατί θα αισθανόμουν ότι θα ήταν πραγματικά άδικο κάποιος που μπορεί να ερευνήσει, μπορεί να επιλέξει να, τους, να χρησιμοποιεί τους κανόνες όπως αυτός θέλει και να οργανώνεται με διαφορετικό τρόπο. Φυσικά μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, αλλά όχι εις βάρος των υπολείπων. Εγώ αν ήμουν μια μικρή επιχείρηση, εφόσον έχω πληρώσει το φόρο που καλούμε να πληρώσω, ε, ε, θα νιώσω ότι θίγομαι που δεν μπορώ να οργανηθώ σε τρεις διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Αυτοί οι οποίοι μας ακούνε σήμερα ε, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ε, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται κάποιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι εις βάρος των υπολείπων που δεν μπορούν να οργανώσουν ε, τα θέματα τους αυτά με τον ίδιο τρόπο. Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες, θα συνεχιστούν οι έρευνες, θα τεκμηριωθούν οι έρευνες και στο τέλος θα δούμε ε, στα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε έτσι ώστε ο κόσμος να έχει ε, πίστη, εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τώρα εκ μέρους Επιτροπής της Εσωτερικής Αγοράς, Σοσιαλιστική Ομάδα, Μαχκ Ταχαμπίλα. Κύριε Επίτροπε, η ψηφιακή εσωτερική αγορά κινδυνεύει από, τον υπερβολικό κατακαιρματισμό της αγοράς και την κατάχρηση δεσποζουσών θέσεων. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε μια αυστηρή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για τον, για ανταγωνισμό ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στη διαγραμμική τεχνολογία και προστασία του καταναλωτή και επίσης μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις αγοράς από μηχανές αναζήτησης στο ίντερνετ που ε, συσσωρεύουν, συλλέγουν, αποθηκεύουν και πολλές φορές για λόγους καθαρά ε, εμπορικούς και πάντως καταχρηστικά εκμεταλλεύονται τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών. Ε, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αν τελικά ψηφιστείτε στη θέση του Επιτρόπου θα είσαστε και πάρα πολύ τυχεροί γιατί έρθετε να ζήσετε στις Βρυξέλλες που είναι η χώρα της καλύτερης σοκολάτας στον κόσμο. I'm going to make my own Αυτό θα το διερευνήσω μόνη μου. Oh, ένα από τα συζητήματα που είναι από τα πιο προβεβλημένα στο νέο κανονισμό για τις γενικές ε, ε, παρεκκλήσεις είναι η πρόσβαση στην υποστήριξη για την ευρυζωνική τεχνολογία εκεί όπου δεν μπορεί να αρκέσει η αγορά. Το να υποσχεθούμε ότι θα έχει ο καθένας την ίδια πρόσβαση στο διαδίκτυο θα ήταν υπερβολικά ε, τολμηρό, γιατί γνωρίζουμε ότι σε ορισμένε περιφέρειε, ε, περιοχέ, χώρε, θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ε, σταθερή πρόσβαση στο ίντερνετ όπως θα θέλαμε όλοι να υπάρχει. Ο νέος λοιπόν αυτός κανονισμός για τις γενικές παρεκκλήσεις δίνει στα κράτη-μέλη νέες δυνατότητες ώστε να μπορούν τα κράτη να εξασφαλίζουν ότι ένας πολίτης που ζει σε μια πιο απομακρυσμένη περιοχή όπου δεν είναι σε θέση η αγορά να προσφέρει επαρκείς ε, υπηρεσίες να μπορεί να τις έχει ο πολίτης τις υπηρεσίες αυτές. Και αυτή είναι η παρέκκληση με μέλημα των καταναλωτή. Γιατί όλο και περισσότερε υπηρεσίε προσφέρονται μέσω του διαδικτύου, όχι μόνο ιδιωτικού τύπου, αλλά και δημοσίου. σχέσει με τις ε, αρχές για παραδείγμα τη ενημέρωση για μετακόμιση, ενημέρωση στο σύστημα υγείας ότι αλλάζουμε γιατρό και το καθεξής. Είναι πράγματα τα οποία σημαίνουν πως χρειάζεται καθνής να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και γι' αυτό νομίζω ότι οι νέοι κανονισμοί που θα έχουν από αυτή την έννοια, από αυτή την άποψη μεγάλη σημασία. Και στο ε, διαδίκτυο διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι η αγορά από την χάνει να, να ρυθμίσει τα προβλήματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπορούμε να παρέμβουμε και να προσφέρουμε υπηρεσία για τον καταναλωτή. Και κάτι το οποίο θα ήθελα να αποκομίσουν οι εκροατές που παρακολουθούν την ε, συζήτηση είναι ότι πρέπει και το Κοινοβούλιο να επιμείνει εφόσον εγκριθεί, όποιος εγκριθεί στη θέση του ε, Επιτρόπου Ανταγωνισμού θα πρέπει να έχει ισχυρό χαρτοφυλάκιο στα θέματα το, της ψηφιακής αγοράς. Όπως αντίστοιχα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην δυνατότητα να απαγορεύει κανείς την εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Η Βίκη Φόρ τώρα από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, η πρόεδρος της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ. Η ΙΜΚΟ έχει αναλάβει νέες ευθύνε για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Καταρχήν, για τις πλατφόρμες peer-to-peer, ομοτήμο υπήρξε ε, απαγόρευση ορισμένων υπηρεσιών αυτού του είδους στην Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια είναι η δική σας άποψη για τέτοιες ε, πράξεις οι οποίες ενδεχομένως κατακαιρματίζουν την ενιαία ψηφιακή αγορά πρωτού καν ξε, ξεκινήσει. Επίσης υπηρεσίες όπως το WhatsApp ή το Skype. Πώς εξασφαλίζεται ότι παίρνουν οι αρχικοί επενδυτές κάποια ε, απόδοση στο κεφαλαίο τους, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν δεσπόζα καταχρηστική θέση και οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Και επίσης είναι κατάλληλο το δίκαιο ανταγωνισμού μας για τον ψηφιακό κόσμο ή θα χρειαστείτε νέα εργαλεία στον χώρο αυτό. Ποτέ δεν θα προσπαθούσα να διορθώσω τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων είναι σημαντικό όμως το γεγονός ότι κάποιες από τις ψηφιακές υπηρεσίες διευκολύνουν νέους τρόπους ανταγωνισμού. Αν αυτός ο ανταγωνισμός είναι θεμητός, αν πληρώνουν τους φόρους και τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν, αυτό το θεωρώ θετικό. Και παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές τις ε, προκλήσεις αποτελούν εκπλήξεις για τις ε, εταιρείε του τομέα, αυτό είναι καλό όσο είναι θεμητός και δίκαιος ο ανταγωνισμός. γιατί πολλές φορές οι καινούργιε αυτές εταιρείε ξέρουν τι φόρους πρέπει να πληρώσουν και τους πληρώνουν και τηρούν τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να ισχύει όταν υπάρχουν νέες αγορές οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν λόγω καινοτομία στον τομέα της πληροφορικής και της, του ψηφιακού θεματολογίου. Νομίζω ότι οι κανόνες ανταγωνισμού που έχουμε είναι υγιείς και όσο πιο σύγχρονοι μπορούσαν να είναι. Απλώς εμείς θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ευφυείς και να έχουμε μεγαλύτερη ε, οξυδέρκεια στο πώς παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές. Κάποιες εταιρείε δεν θεωρούν τον εαυτό τους ότι δεν είναι καν ε, εθνικές ή ευρωπαϊκές θεωρούν από τη στιγμή μηδέν ότι είναι παγκόσμιες γιατί η παγκόσμια είναι η αγορά που θέλουν να κατακτήσουν και αυτή είναι η πρόκληση να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις και όχι απλώς να ελκόμαστε από όλα αυτά αλλά να έχουμε μια πλήρη κατανόηση κάποια πράγματα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού, όπως παραδείγματος χάρη συζήτηση για το big data, για τα προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα που συλλέγονται, γιατί όλα αυτά αλλάζουν και την αντιμετώπιση που έχουμε για την αξία που έχουν τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα ουσιαστικά νομίσματος τα προσωπικά δεδομένα ε, πηγή αξία σε ορισμένε από τι πίεσει που χρησιμοποιούμε. Ελπίζω ότι πολλά από αυτά θα μπορέσουμε να τα κάνουμε από κοινού. Ειρήνα Κάρη τώρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ εξεπλάγει λιγάκι με αυτό που είπατε για το για ορισμένε υπηρεσίε στο διαδίκτυο. Ή, τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί οι δημόσιες αρρωγές στην ε, Δανία οδήγησαν σε ένα αύξηση κατά 5% ε, των μισθών των ε, εργαζόμενων στην αυπηγική βιομηχανία. Αυτό όμως οδήγησε στους, ε, στις επιχειρήσεις ναυπήγησης να φέρουν εργαζόμενους από άλλες χώρες κάτω από αποτρόπες συνθήκες εργασίας και πληρωμής. Ως αρμόδια για τον ανταγωνισμό θα πρέπει να είσαστε αρμόδια για τον ανταγωνισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι είναι θεμητός ανταγωνισμός να έρχονται εργαζόμενοι κάτω από αυτές τις συνθήκες και μετά αυτές οι επιχειρήσεις, οι εφοπλιστές, οι ναυπηγικές εταιρείες να παίρνουν επιδοτήσεις για να φέρουν εργαζόμενους κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εγώ δεν νομίζω αυτό δεν είναι, ότι δεν είναι προς όφελος κανενός. Για μένα, λέει η κυρία Βέστογκερ, όταν προετοιμαζόμουν για αυτήν την ακρόαση, το πιο σημαντικό ήταν να προετοιμαστώ για να έχω ένα χαρακτήρα ανεξάρτητο. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι αναπόδραστο για να μπορέσω να είμαι πραγματική επίτροπος ανταγωνισμού, εφόσον φυσικά εγκρίνεται την υποψηφιότητά μου. Πέραν όλων αυτό που θα μπορούσα να έχω κάνει ή να έχω σκεφτεί όταν ήμουνα βουλευτής ή υπουργός στη Δανία, εγώ εδώ πρέπει να αναλάβω μια ευθύνη πολύ διαφορετική εδώ. Γιατί στον πυρήνα της δραστηριότητάς μου είναι ότι δεν θα μπορώ ούτε θα πρέπει να παίρνω εντολές από κανένα, ούτε θα πρέπει να τις ζητώ αυτές τις εντολές. Η ανεξαρτησία στο έργο μου είναι απαραίτητη. Επομένως, δεν με ενδιαφέρει αν ένας μηχανισμός είναι, δα, είναι από, από τη Δανία ή από κάπου αλλού. Με ενδιαφέρεται αν είναι κάτι το οποίο είναι συνάδων με τους κανόνες ή όχι. Υπάρχουν πολλά χρόνια λοιπόν που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα για τον ανταγωνισμό και όλοι οι επίτροποι που έχουν αναλάβει αυτό το έργο έχουν συμμορφωθεί με αυτό το πλαίσιο. Τελευταία ερώτηση από την Κάτια Κάλλας της Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι μια και έχω υπηρετήσει ως δικηγόρος ανταγωνισμού για 40 χρόνια, βλέπω με πολύ αισιοδοξία ότι θα είναι σε καλά χέρια ο ανταγωνισμός στην Επιτροπή. Αλλά έχω μια ερώτηση για την Google από μια άλλη σκοπιά. Κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν από Ευρωπαίους ηγέτες με ανησυχούν. Πρόκειται για σχόλια που λένε ότι για να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την ψηφιακή υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Google θα πρέπει να επιβληθούν ε, παραπάνω, ε, παραπάνω περιορισμοί και ρυθμίσεις στο ίντερνετ, ίσως και υπερβολικές ρυθμίσεις. Ερωτώ λοιπόν πώς θα συνεργαστείτε με τους άλλους συναρμόδιους επιτρόπους ώστε να αντιμετωπίσετε την ε, πολιτική αυτή κάποιων κρατών που μπορεί να στρέφεται και κατά του ανταγωνισμού και θα σημαίνει υπερβολικό έλεγχο στο ίντερνετ. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ω τελευταία ερώτηση νομίζω έρχεται στην κατάλληλη στιγμή και είναι η καταλληλότερη ερώτηση διότι ε, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι αδίποτε έρευνα στηρίζεται σε γεγονότα και πραγματικά περιστατικά. Όχι σε συναισθήματα, όχι σε πολιτικές ιδεολογίες, όχι σε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Γιατί αυτό είναι ο μόνος, ο μόνος τρόπος να τηρήσουμε τη βασική αυτή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το κράτος δικαίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν κάνουμε μια έρευνα, όταν κάνουμε μια υπόθεση, την ερευνούμε με βάση τα πραγματικά περιστατικά, με αντίληψη του τι σημαίνει η αγορά, τι κάνει η αγορά και με ε, τους κανόνες υπόψη που πρόκειται να εφαρμόσουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταθεί και στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. Και είναι πολύ σημαντικό διότι τα δικαστήρια είναι αυτά τα οποία εν τέλει φροντίζουν να βρουν και να δώσουν τις λεπτές αυτές τι ισορροπίες που χρειάζονται. Έχει τεράστιες εκτελεστικές εξουσίες ως προς τον ανταγωνισμό η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, εάν κανείς προσφύγει στα δικαστήρια μετά την ε, απόφαση της Επιτροπής ε, στο θέμα του ανταγωνισμού, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή να μην ανατραπεί. Και γι' αυτό εγώ θέλω να φροντίζω πάντα να βεβαιωνόμαι ότι έχουμε τηρήσει κάθε διάταξη του χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ότι όλοι οι κανόνες τηρούνται σωστά, ώστε και να ε, εξασφαλίζουμε την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την επιβολή τους με έναν τρόπο ουδέτερο, στηριζόμενο σε πραγματικά περιστατικά και αδέκαστο. Και ελπίζω να έχετε δίκιο, γιατί ακριβώς αυτό φοβόμουν. Άνθρωποι που για 20, 30, 40 χρόνια δουλεύουν στον τομέα αυτών, Φοβόμουν ότι θα μου λέγανε ότι δεν είμαι επαρκής. Ε, με ενθαρρύνουν πολύ λοιπόν τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις τους. Και τώρα θα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά στην ε, υποψήφια επίτροπο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω εφόσον ε, εσείς ασχολείστε και με τα θέματα ε, του, ειδικά με τα θέματα του ανταγωνισμού στην ΙΜΚΟ και σας θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι από όλε τι ερωτήσεις ε, ένα πράγμα βγήκε σαν μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον ανταγωνισμό ένα ουδέτερο ε, δίκαιο τρόπο εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα ε, δόθηκε και πώς ε, η εφαρμογή του ανταγωνισμού θα διευκολύνει και θα βοηθήσει και άλλους τομείς οικονομικούς και πολιτικούς. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας σε κάποια από τα θέματα ίσως δεν στάθηκα πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ελπίζω να επανέλθουμε, να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να εκτιμήσατε ότι προσπάθησα να σας δείξω το ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές τις οποίες πρεσβεύω και θα είναι η βάση της συνεργασίας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το μήνυμα από την συνάντηση αυτή, από την ακρόαση αυτή, είναι η δυνατότητα και η πίστη που έχουμε στον ανταγωνισμό που θα βοηθήσει τις περισσότερες επενδύσεις, την απασχόληση ε, και τις θέσεις απασχόλησης κυρίως. Ε, όλοι συνειδητοποιούμε επίσης το τι σημαίνει ε, η ψηφιακή οικονομία για τους πολίτες και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός και όχι κυρίαρχη θέση. Διότι είναι σημαντικό για τον καταναλωτή και για τον υπολογιστή λέει η υποψηφία επίτροπος. κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου εδώ έμαθα πάρα πολλά αρχικά. Μιλάμε για διάφορα αρχικά σε διάφορους τομείς. Και μετά έπεσα σε κάτι ρυθμίσεις για τον τρόπο με τον οποίο συναρμολογούνται τα παράθυρα και αναρωτήθηκα τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό αποφάσεις για την συναρμολόγηση των παραθύρων. Ε, αφορούσε τα παράθυρα. Γιατί η παραγωγή ακριβώς ε, τέτοιου είδους κουφωμάτων ε, πράγματι ε, ήθελαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και πράγματι υπήρξε μία απόφαση για τα κουφώματα των παραθύρων. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εταιρείες προσπάθησαν ιδιαίτερα για να προωθήσουν αυτές τις απόψεις. Καταλαβαίνετε ότι μετά από μια τέτοια εμπειρία πώς ένιωσα. Αυτό το οποίο με βοήθησε πάντως είναι ότι η συνεργασία με σας ε, ε, πράγματι μπορεί να πάρει πολύ σημαντική, σημαντικό ρόλο. και μπορούμε να πετύχουμε πολλά συνεργαζόμενοι και επίσημα και ανεπίσημα Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως ε, είπα επανειλημμένα ε, θα προσπαθήσω να πάρω μέρος σε αυτή τη μορφή συνεργασίας. Είμαι κόρη ιερέων στην εκκλησία της χώρας μου και μία από τις βασικές τους αρετές ήταν ότι καλωσόριζαν πάντα όσους έμπαιναν στην εκκλησία. Αντί να λένε άσχημα πράγματα για αυτούς που δεν έμπαιναν στην εκκλησία. Και γι' αυτό <laughs> καλωσορίζω όλους εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Because I, I think it shows the dedication, which is actually and truly there. Αυτό δείχνει ακριβώς την αφοσίωσή σας στην υπόθεση αυτή. Και ελπίζω να είμαι ξεκάθαρη, θέλω να ευχαριστήσω τη διερμηνία, ελπίζω να διευκόλυναν αυτά τα οποία είπα την κατανόησή τους. Αγαπητά μέλη λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ Μάργαρετ Βέστακερ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την υπομονή. Τελειώνει εδώ η συνεδρίαση και σε 30 λεπτά έχουμε την αξιολόγησή μας και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστώ, πέρα συνεδριάσεως.